Euh, Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αρκετά φορτωμένη η σημερινή μας ημερήσια διάταξη, γι' αυτό ας αρχίσουμε αμέσως. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά της συνεδρίας 1 Φεβρουαρίου, εγκρίνονται. Σήμερα έχουμε τέσσερα σημεία στην ημερήσια διάταξη, δύο από τα οποία αφορούν τα Βαλκάνια με τη μη στρατιωτική αποστολή Γιούλεξ στο Κοφισιφοπέδιο και την αστυνομική αποστολή στη Βονζία Ζεγοβίνη και μετά έχουμε την έκθεση Γκουαλτιέρη στις 11.30 ο κύριος Ποπόφσκι ε, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της, ε, εξωτερικής, της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης θα μας μιλήσει για τη Λιβύη. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρώτα απ' όλα τον διοικητή πολιτικών δράσεων Κόμπενχάουερ, τον κύριο Μπούντο Μαρνιάκ, επικεφαλής αντιπροσωπείας της ε, Γιούλεξ στο Κωσυφοπέδι και τον κύριο Στέφαν Φέλερ της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. Όπως ξέρετε, σήμερα μας παρα... απασχολούν ιδιαίτερα τα θέματα ασφαλείας που αφορούν τη Λιβύη. Μετά από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Παρασκευής θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε για το θέμα αυτό τον κύριο Ποπόφσκι. Θελήσαμε παρόλα αυτά να παραμείνει η μερίσια διάταξη έτσι όπως είχε οργανωθεί για να συζητήσουμε για τα Βαλκάνια, δεδομένου ότι οι δύο μη στρατιωτικές αποστολές στα Βαλκάνια είναι πάρα πολύ σημαντικές από πολιτικής πλευράς και από ε, όσον αφορά την άτομα που συμμετέχουν. Πρόκειται για αποστολές οι οποίες είναι πρωταρχικής σημασίας για να κατοπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και να μπορέσει να παγιωθεί το κράτος δικαίου στο κοσυφοπαίδιο. Στην ε, Γιούλεξ έχουμε ε, γεγονότα επικαιρότητα πάρα πολύ σημαντικά. Μετά από την έκθεση Μάρτη για την εμπορία ανθρωπίνων οργάνων στο Κωσυφοπαίδιο και την Αλβανία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν όντως η ΛΕΞ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, όπως είπε και ο κύριος Μάρτη, για την προστασία των μαρτύρων. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας και με μεγάλη ευχαρίστηση θα ακούσουμε τον επικεφαλής της αποστολής για το θέμα αυτό. Εκτός από την έκθεση Μάρτη, η οποία όντως είναι επίκαιρη και σημαντικότατη, θα πρέπει να κάνουμε και αξιολόγηση της ε, αποστολής ΕΛΕΞΕ σε όλες τις πτυχές της, για όλα τα θέματα επικαιρότητα στην Πρίστινα, τις δίκες. Επίσης, να μας πείτε από θέματα στρατηγικής πώς πιστεύετε ότι για θέματα δικαιοσύνης και θέματα τελωνιακά αναπτύσσεται η δική σας δύναμη. Θα κάνουμε λοιπόν μία πλήρη εξέταση της όλης αποστολής της Γιούλεξ πέραν τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά τα συμπεράσματα της ε, έκθεσης Μάρτη. Ο προκάτοχός σας είχε έρθει στην Επιτροπή μας πριν από 6 μήνες. Χαιρόμεθα που έχουμε λοιπόν ε, και πάλι μια νέα συνάντηση μαζί σας. Πριν, ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, δίδω πρώτα το λόγο στον κύριο Κλόπενχαουρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και στον κύριο Ντεμαρνάκ. Ευχαριστώ. Είναι τέταρτη φορά κύριε Πρόεδρε που συμμετέχω στις συζητήσεις της Επιτροπής σας και χαίρομαι ιδιαίτερα. Όντω είναι μεγάλο μου πλέον προνόμιο να βρίσκομαι εδώ μαζί σα σήμερα για να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα πολιτικών δράσεων στα Βαλκάνια. Οι δράσεις λοιπόν αυτές, οι ενέργειες αυτές αποτυπώνουν τη δεσμεύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιφέρεια όπου υπάρχει ιδιαίτερη ευθύνη και όπου έχει χρησιμοποιηθεί όλη η ομάδα των μέσων που υπάρχουν. Θα σας αναφέρουμε, θα αναφέρει ο κύριος Τσέιντ ε, τις ε, δραστηριότητες και των δύο ομάδων. Θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας για κάποια βασικά ζητήματα, τα οποία είναι ουσιώδη για την καλή λειτουργία και την επιτυχία και του ULAX και του e UPM. Ο Ξαβιέ και ο Στέφαν θα σας κάνουν μια ενημέρωση για την κατάσταση στην περιοχή και για τις σχετικές δράσεις που έχουν αναλυφθεί. Ένα πρώτο θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το οποίο ο Πρόεδρος ήδη ανέφερε είναι η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Τικμαχτή. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει κάποιες αιτιάσεις τις οποίες λαμβάνει πολύ σοβαρά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την δεκαετία του 90, τέλη της δεκαετίας 90 για κάποια εγκλήματα τα οποία έλεγαν χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα εξετάσει αυτά, όπως είπα, με ενδελέχεια και έχουν γίνει πολλές ε, εικασίες στα διεθνή φόρα για την Ιουλέξ και για την ικανότητά της να παρακολουθήσει και να συνεχίσει την έκθεση Μάρτη. Να είμαι σαφής, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν αμφιβολίες για το θέμα αυτό. Η Ιουλέξ έχει την κατάλληλη εντολή για να ερευνήσει τα ζητήματα αυτά συμπεριλαμβανομένων και των συνεπειών στην περιφέρεια. Και ο Ξχαβιέ θα επισέλθει σε λεπτομέρειες για τις ε, διακανονισμό που έχει κάνει. Θα ήθελα επίσης να καταστάσω σαφές ότι πρόκειται για μία μόνο από τις πολλές υποθέσεις που ερευνάει η Γιούλεξ Πράγματι, Πρόκειται για έναν από τους βασικούς μας στόχους. Θέλουμε να μεταφέρουμε τις ε, έρευνες σε ευαίσθητες υποθέσεις ε, και να τις καταστήσουμε, ε, να δώσουμε μάλλον βάση για να υπάρχουν έρευνες από εισαγγελικέ αρχές. Αυτές λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος της ULEX και επίσης να υπάρχει έντονο αποτύπωμα της δράσης μας στο σύγχρονο κοσυφοπαίδιο με επίκεντρο τις εγκληματικές δράσεις και επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε αυτούς τους δύο στόχους συνεχίζοντας και τις ε, υπόλοιπες δραστηριότητε μας. Θα ήθελα να περάσω τώρα στην Βοσνία Σεγοβίνη εν συντομία σε ό,τι αφορά το EUPM εξακολουθούν να υπάρχουν α, ε, ε, κατηγορίες και χρειάζονται καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ε, ε, προκλήσεις αυτές χρειάζεται διαφάνεια στο σύστημα εφαρμογής του νόμου στην Ποσνία Ζεγοβίνη και θα σας ενημερώσουμε πώς σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε την υπόλοιπη εντολή μας φέτος για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Τέλος, και αυτό το λέω πάντα, αλλά το επαναλαμβάνω επειδή ακριβώ είναι σημαντικό για να τα πετύχουμε όλα αυτά, χρειαζόμαστε την πολιτική σας υποστήριξη. Και την υλική υποστήριξη και πολιτική υποστήριξη των κυβερνήσεων. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό και, κατά περίπτωση, πιο μεγάλη ευελιξία. Θα πρέπει να εισαχθεί περισσότερη ευελιξία για να έχουμε πιο πολλούς συμβασιούχους σε αποστολές όταν δεν έχουμε αποσπασμένο προσωπικό. Σε μια φάση όπου η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και οι πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις ενδεχομένως να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα Βαλκάνια, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει να μείνει ατελείωτο το έργο της ε, στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν υπολογίζω στην υποστήριξή σας και των εθνικών κυβερνήσεων για να ολοκληρώσουμε τη σημαντική μας δράση στα Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Για να είναι εύληπτα, εύληπτες οι συζητήσεις, ε, θα ήθελα παρότι έχουμε δύο αποστολές για το ίδιο θέμα, για τα Βαλκάνια δηλαδή, να ξεχωρίσουμε τις συζητήσεις. Καταρχάς να μιλήσουμε για τη ULEX, ε, μετά να συζητήσουμε για το Κοσφοπέδιο και μετά για τη Βοσνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως επικεφαλής ε, της αποστολής για την ε, δημιουργία κράτους δικαίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω σήμερα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κοσφοπέδιο. Θα εστιάσω την παρέμβασή μου στην έκθεση που υπάρχει και στις προτεραιότητες για την αποστολή μας. Από τη στιγμή που ανέλαβα από, το, από τον Ιβντο και Αμαμπό τον Οκτώβριο του 2010. Θα ήθελα καταρχάς να περιγράψω συντομία την κατάσταση επιτόπου. Η συνολική κατάσταση στο Κοσφοπέδιο ε, είναι ήρεμη σε μια περίοδο ε, σημαντικών πολιτικών ε, ζυμώσεων, όπως θα γνωρίζουν πολλοί από εσά. Η πρόσφατη δημιουργία μιας νέας πολιτικής ηγεσία του Κωσυφοπεδίου θα μας επιτρέψει να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα του κράτους δικαίου. Οι, τρει τρεις Υπουργοί Εσωτερικών Δικαιοσύνης και Οικονομικών ε, μου είναι γνωστοί και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί με επικοδομητικό τρόπο. Με, την, τη δημιουργία τώρα ε, θεσμικής ηγεσία μπορούμε να θέσουμε κοινού στόχους σε στενή συνεργασία και συντονισμό ε, για το, την προετοιμασία των δύο εκθέσεων ε, του 2011. Με αυτόν τον ε, τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε κοινέ προσπάθειες ούτως ώστε να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και κυρίως για να υπάρξει ε, συνεκτικότητα στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες στο κοσφοπέδιο. Τούτου λεχθέντος. Ε, Βεβαίω η κατάσταση είναι ήρεμη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σημάδια ανησυχίας και ε, προβλημάτων. Υπάρχουν κίνδυνοι α, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του κοσφοπεδίου υπάρχει η αντίληψη ότι μεγαλώνει η απομονωσή του και υπάρχουν και πολλές προσδοκίες από το καθεστώς απελευθέρωσης της υποχρέωσης θεωρήσεων. Το βόρειο τμήμα του Κοσφοπεδίου ε, έχει εντάσεις και ελπίζω ειλικρινά ότι ο διάλογος μεταξύ της Πριστίνας και του Βελιγραδίου που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όπως ξέρετε, θα φέρει τις δύο κοινότητες πιο κοντά τη μία στην άλλη σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Η ULEX είναι αποφασισμένη να βοηθήσει όσο μπορεί για να υποστηρίξει τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ε, τώρα πάω στην έκθεση του γερουσιαστή Dick Martin. Όπως ξέρετε, η αποστολή έχει λάβει σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς του κυρίου Μάρτι, όπως εμφανίζονται στην έκθεσή του. Πάρα αυτά, μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος από το Συμβούλιο της Ευρώπης βάσει της έκθεσης, η Γιούλεξ ξεκίνησε μία προκαταρτική έρευνα ε, για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς της έκθεσης αυτής. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση της έρευνας δεν υπάρχουν υποψίες ε, και ύποπτοι, ύποπτοι μάλλον. Θα ήθελα να πω ότι οι εισαγγελίες της Γιούλεξ έχουν δικαιοδοσία για να διερευνήσουν τους ε, ισχυρισμούς του κ. Μάρτη τις επόμενες εβδομάδες η Γιούλεξ ε, θα κάνει τα εξής πράγματα σε σχέση με την έκθεση αυτή. Η αποστολή θα επιλέξει ε, το κατάλληλο προσωπικό που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με τους ισχυρισμούς αυτούς. Θα υπάρξει υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί, το προσωπικό αυτό, να λειτουργήσει μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο θα καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχύσουμε την προστασία των μαρτύρων που συμπεριλαμβάνει και πρόγραμμα επανεγκατάστασης μαρτύρων. Η συνεργασία με τέρους και στο Βελιγράδι και στα Τύρανα μέχρι στιγμής λειτουργήσε ικανοποιητικά και θα συνεχιστεί ε, όπως μέχρι σήμερα. Μετά την... Ε, θα υπάρξει μεγάλη προσοχή από τη Γιούλεξ ε, στο follow-up της έκθεσης Μάρτη. Θα ήθελα να σας πω ότι οι δύο βασικές προτεραιότητές μας είναι οι εξή. Τις έχω εντοπίσει από τη στιγμή που ανέλαβα αυτή τη θέση βέβαια. Πρώτον, είναι το βόρειο τμήμα του Κοσφοπεδίου, όπου η προτεραιότητά μου είναι να διατηρήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον. Η προσέγγιση μου ε, για να εφαρμοστεί αυτή η προτεραιότητα είναι διτή. Είμαστε σε μια φάση επέκταση του αποτυπώματό μα και ενίσχυση της παρουσίας μας στο βόρειο τμήμα του Κοσφοπεδίου και ταυτόχρονα εφαρμόζουμε ε, το δίκαιο. Ε, καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο η Γιούλεξ θα καταλάβει καλύτερα την κατάσταση και θα διευκολυνθεί η αποδοχή μας από τον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ανταλλαγή και ε, τακτικές επαφές μεταξύ των μελών τη αποστολή και τη τοπική ηγεσία, ούτω ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσει μεταξύ μα. Επιπλέον, πέρα από το, το σημαντικό διοικητικό βήμα, θα δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και του πληθυσμού, καταπολεμώντας τις εγκληματικές δομές που ενεργοποιούνται στο βορρά. Αυτές οι διοκτικές προσπάθειες ε, γίνονται στο κοσφοπέδιο και θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ομάδες τις ε, διακοινωτικές ε, που λειτουργούν ένθεν και ένθεν του ποταμού Ήμπερ. Η πρώτη σημαντική επιχείρηση ξεκίνησε το Φεβρουάριο με την πλήρη υποστήριξη της K4 και θα υπάρξουν και νέες επιχειρήσεις στο εγγύς μέλλον. Μετά την επίσκεψή μου στο Βελιγράδι, επίσης περιμένω να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση από τις ε, σερβικές αρχές για να προβούμε σε κάποιες έρευνες. Η δεύτερη σημαντική μου προτεραιότητα είναι μια μεγάλη δέσμευση να διεκπαιρεώσουμε σημαντικές υποθέσεις εναντίον περιπτώσεων οργανωμένου εγκλήματος και ε, διαφθοράς. Γνωρίζω ότι την αποστολή θα την κρίνουν με βάση τα επιτεύγματά της και σε αυτό το τομέα. Και είμαι απόλυτα αποφασισμένος τα λόγια αυτά να τα κάνω πράξη. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, των εγκλημάτων πολέμου και της διαφθοράς είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και σε ορισμένες περιπτώσεις σκοπεύω να συνεργαστώ εκ του σύγκης με τους τοπικούς φορείς και όλο και, μάλιστα και όλο και πιο στενά. Το 2010 ε, χαρακτηρίστηκε από πολλές ε, περίπλοκες και ευαίσθητες ε, έρευνες από τους εισαγγελεί τη Γιούλεξ. Είμαι πεπισμένο ότι αυτή η σκληρή δουλειά θα δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα υπάρξουν διώξει και θα υπάρξουν και περιπτώσει που θα φτάσουν στα δικαστήρια μέσα στο 2011. Τους επόμενους μήνες η προτεραιότητα θα δοθεί στο οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο να βελτιώσουμε το κράτο δικαίου στο κοσφοπέδιο, αλλά να βελτιώσουμε και την ασφάλεια και για τα κράτη-μέλη. Είμαι πεπισμένος ότι οι αρχέ του Κοσφοπεδίου έχουν την ικανότητα και τη δέσμευση, ιδίω η αστυνομία του Κοσφοπεδίου, μαζί με τη Γιούλεξ να δώσουν αποτελέσματα, οι προσπάθειέ να δώσουν αποτελέσματα σε αυτού του τομεί. Τέλο, θέλω να τονίσω τη σημασία να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδο των αρχών του Κοσφοπεδίου καταγράφεται και σημειώνεται σωστά. Η Γιούλεξ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ικανότητα ανάληψης περισσότερων ευθυνών θα λογοδοτήσω λοιπόν στα κράτη-μέλη σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που θα σημειώσουν οι τοπικές αρχές και οι δραστηριότητε τη Αποστολή θα ξεκαθαρίζουν τις προσπάθειες των αρχών του Κωσυφοπεδίου. Τον επόμενο χρόνο πιστεύω ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ενισχύσουν το κράτο δικαίου στο Κωσυφοπέδιο. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Euh, ευχαριστώ. Διάφοροι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Έχω ένα ερώτημα από πλευράς μου για την εντολή. Μετά την έκθεση Μάρτη. Εισαγωγικά αναφέρατε και εσείς κύριε Κλωμεχάρο, αλλά και εσείς ότι η Γιούλεξ έχει την ικανότητα να προβεί σε αυτές τις έρευνες και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το ερώτημα επανέρχεται συνέχεια. Έχετε το δυναμικό το νομικό δυναμικό και έχετε και το δυναμικό στην πράξη να κάνετε αυτές τις ε, έρευνες κυρίως στην Αλβανία, γιατί την αναφέρατε και αυτή η χώρα, αλλά και πέρα από την Αλβανία, σε περίπτωση που κάποιοι εντολοδότες ή κάποιοι δικαιούχοι από, αυτή την, από αυτό το λαθρεμπόριο ε, βρίσκονται σε άλλες χώρες ε, και χώρες μάλιστα εκτός Ευρώπης. Η Γιούλεξ έχει το δυναμικό για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, έχει αυτή την εντολή. Δεύτερο ερώτημα. Ε, για τους α, ε, αγνοούμενους. Έχουμε 1.800 ε, αγνοούμενους, 1.400 Κωσοβάρους, Αλβανούς και 400 Σέρβους. Ανησυχούμε πολύ για την μοίρα τους. Είναι σημαντικό αυτό για τη διαδικασία συμφιλίωσης. Και θα ήθελα να μου πείτε αν η Ulex ε, παίζει, μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο εδώ. Πέρυσι επίσης, όταν ε, ήρθε εδώ ο προκάτοχός σας, είχαμε αναβάλει την ε, πρώτη μας σύνοδο, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη επιχείρηση στην Πριστίνα, για να εντοπιστούν περιπτώσεις διαφθοράς υψηλών αξιωματούχων. Μας είχατε πει ότι θα έχετε γρήγορα αποτελέσματα τότε. Είχατε, ξεκινήσει, τώρα είμαστε ένα χρόνο μετά από αυτή την ε, θεαματική επιχείρηση. Θα ήθελα να μου πείτε αν τα αποτελέσματα που μας υποσχεθήκατε θα υπάρξουν τελικά, γιατί δεν, έχουμε, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Είναι σημαντικό νομίζω μια και δόθηκαν σημαντικά πολιτικά μηνύματα τότε, να δούμε τώρα σήμερα, ένα χρόνο μετά, αν υπάρχουν ε, πραγματικά αποτελέσματα. Τώρα η κυρία Λούνατσεκ που είναι η συγγήτρια του Κοσφοπεδίου, για το Κοσφοπέδιο. Χαίρετε κύριε Κλάπενχάουερ, κύριε Ντεμανιάκ. Στον κύριο Μποντεμανιάκ θα ήθελα να πω ότι την... έρχεστε για πρώτη φορά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και αρχίζοντας θα ήθελα να πω το εξής. Δυστυχώς Πολλές φορές έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά και παρά το γεγονός ότι έκανα κάποιες επικρίσεις πριν να σας γνωρίσω, δηλαδή είπα ότι και πάλι υπάρχει στρατιωτικός επικεφαλής μίας μη στρατιωτικής αποστολής, πρέπει να πω ότι είστε κάποιος ο οποίος έχει ανοιχτές ιδέες και ευθύς εξ αρχής το καταστηριό. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θίξατε και θα ήθελα να αναφέρω κάποια λεπτομεριακό. Όπως είπε και ο κύριος Ντόνζαν στην τελευταία παρατήρησή του, η καταπολέμηση της διαφθοράς, μεγάλη υπόθεση. Η τελευταία περίπτωση άρχισε, όπως ξέρετε, πέρσι τον Απρίλιο. Ξέρετε πώς αισθάνονται οι διάφοροι. Το μεγάλο ψάρι θα το πιάσει τελικά η Γιούλεξ για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις για το αν πιάστηκε αυτό το μεγάλο ψάρι και έχουν υπάρξει και διάφορες επικρίσεις επί του θέματος. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα. Πότε θα περιμένουμε εκδίκες τέτοιου είδους υποθέσεων. Τώρα, η υπόθεση της έκθεσης Μάρτη. Στο Στρασβούργο, ο κύριος Μάρτη, σε μία συνεδρίαση και κλεισμένο το θηρόν της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, συμμετείχε σε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να φέρω κάποια θέματα και κ. κύριο Χάουρ, θίξατε. Όντως, τα κράτη-μέλη δεν δίδουν κυρίως το κατάλληλο δικαστικό προσωπικό για να βοηθήσουν την αποστολή σας όπως θα έπρεπε να γίνει. Είπατε ότι έχετε αρχίσει κάποιες έρευνες και τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσετε με το θέμα της προστασίας με την κατάσταση των μαρτύρων. Τι χρειάζεστε από τα κρατημέλη, πόσα περαιτέρω άτομα, εισαγγελείς ή άλλο δικαστικό προσωπικό χρειάζεστε, όχι μόνο για τις υποθέσεις ε, τις οποίες πραγματεύεται η έκθεση Μάρτη, αλλά γενικότερα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την αποστολή σας και την εντολή σας. Το επόμενο θέμα είναι ότι παρουσιάστηκε η ιδέα ενδεχομένω με τη συνδρομή της Ulex να γίνουν ίσω κάποιες δίκε δίκες εκτός κοσυφοπεδίου, σε ουδέτερο διότι υπάρχουν φόβοι ότι στην ε, περιοχή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα προστασίας των μαρτύρων, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Τι έχετε να πείτε για το θέμα αυτό. Τώρα, για το Βορρά, είπατε εσείς ε, ότι θέλετε να παραμείνει ε, το όλο κλίμα που θα δημιουργηθεί κυρίως στο βορρά σταθερό. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει ε, παρά μόνο ελάχιστη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Είπετε ότι θέλετε να μπορέσετε να έχετε κλίμα εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί με την τοπική εκεί αυτοδιοίκηση. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Ο διάλογος επίσης μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας πιστεύετε ότι είναι κάποια οδός πρόοδου κάποιος τρόπος θα βοηθήσει την όλη κατάσταση να εξελιχθεί θετικά. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν, πρόεδρος Επιτροπής για την ατελική ευρωπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δύο-τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τους τρεις κυρίους. Πραγματικά εκτιμούμε την εργασία που επιτελείται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μαζί σας αυτή την ανταλλαγή απόψεως. Επίσης, εκτιμώ την πάρα πολύ πραγματιστική άποψή σας για το τι ακριβώς διαμείβεται στην περιοχή αυτή της οποίας έχετε την ευθύνη. Όπως και προείσχαμε με την προηγούμενη εβδομάδα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ντικ Μάρτι διαφορετική από τη σημερινή ίσως. Το ερώτημά μας στον κύριο Ντε Μαρνιάκ είναι ότι στις 28 Ιανουαρίου έκανε μια δήλωση Γιούλοξ και είπε ότι έχει την δυνατότητα, την δικαιοδοσία και την πραγματογνωσύνη που χρειάζεται για να παρακολουθεί τέτοιου είδους ε, υποθέσεις στον δικαστικό τομέα θέμα μου είναι και εμένα πώς μπορούν να σας βοηθήσουν ε, όπως ελέγχθη τα ε, κράτη-μέλη και εγώ προσθέτω πώς μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κύριος Μαρτί βοηθά. Δεύτερον, τι συμβαίνει με την υπόθεση Θόρτερ Λίμαϊ. Ευχαριστώ κυρία Πακ. Σας ευχαριστώ κύριε που βρίσκεστε εδώ και έχουμε την τιμή να έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και να συζητήσουμε για θέματα Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Τέσσερις ερωτήσεις έχω. Η πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα... Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε πόσες περιπτώσεις ε, που έχει επιλύσει η ούνμικ και που είχε αλλάσει, αφήσει μάλλον ε, η ουνμίκ έχει καταφέρει η Γιούλεξ να τις ε, λύσει, να τις ε, φέρει σε μια φάση απόφασης. Δεύτερον, κατά την αλλαγή των πρώην υπαλλήλων της ουνμίκ σε κομματικά, σε κομματικούς κύκλους, θεωρείται ότι αυτό είναι προβληματικό και υπάρχουν σχετικές διώξεις. Ο κύριος Μάρτιν, τρίτον, στις δηλώσεις του είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ ιδιαίτερα. Όχι, δεν συμφωνώ με όλα, αλλά με αυτό συμφωνώ. Ότι για την δίωξη κάθε δεύτερης περίπτωσης διαφθοράς ή για αυτές τις ε, κατηγορίες για την εμπορία οργάνων θα χρειαζόμαστε υπαλλήλου τη ε, Ulex οι οποίοι θα ήταν στο Κωσυφοπέδιο για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί δεν έχει νόημα να μπει ε, ένα υπάλληλο μέσα στην όλη κατάσταση και μετά λόγω κινητικότητα να αναγκαστεί να φύγει και να έρθει ένα καινούριο. Θεωρώ ότι σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις θα πρέπει να βρούμε μια δυνατότητα για κάποια άτομα τα οποία έχουν μπει μέσα στην υπόθεση να μείνουν μέχρι ότου ολοκληρωθεί η υπόθεση. Τελευταία ερώτηση. Το ανέφερε και ο Αρνό το πρόβλημα του μέχρι πού φτάνει η εξουσία της ε, ε, στην Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζω, ε, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει και να συνεργαστεί απόλυτα. Αυτή την προσφορά μπορείτε να την αποδεχτείτε. Καν. Ευχαριστώ. Merci, Madame Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις για τον κύριο Κλόμπενχάουαρ και μία ερώτηση για τον κύριο Ντεμαρνιάκ. Κύριε Κλόμπονάουερ, πρώτη ερώτηση για τον στόχο της πολιτικής αποστολής που λέγει το 2010. Μία αξιολόγηση θα ήθελα να μου κάνετε για το πώς έχει η κατάσταση σήμερα και αν θεωρείτε ότι είναι δέουσα μία διαδικασία follow-up και υπό ποια μορφή. Δεύτερη ερώτηση, η συμμετοχή στα Βαλκάνια δεδομένων και των εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Ξέρω για την αφαίρεση των ε, ναρκών. Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες, αλλά αν θα μπορούσατε να μας ε, πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση στη Βοσνία Ριζαγοβίνη και στο Κωσυφοπίδιο, γιατί ξέρουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές νάρκες στις νοριακές περιοχές ε, που προκαλούν ασφαλώς πολλά προβλήματα. Ερωτώ λοιπόν και τον κύριο Τερμαρνιάκ. Δεν μιλήσατε για το βασικό θέμα, λυπάμαι, το οποίο ανακύπτει από την έκθεση Μαρτή που αφορά την προστασία των μαρτύρων γιατί μας παρουσίασε κάποιες τρομακτικά αριθμητικά στοιχεία δολοφονιών στην έκθεση του Στρασβούργο. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το βασικότατο αυτό πρόβλημα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν είναι πολύ καλά οργανωμένη η έρευνα, αν τελικά ο κόσμος δεν προστατεύεται, πολύ απλά δεν θα βγει να μιλήσει. Λόγω της ιστορίας της ε, περιοχής. Εξηγήστε μας λοιπόν, αν θέλετε, ποια είναι η στρατηγική σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρλάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τις ε, δηλώσεις του κυρίου Κλόμπενχάουερ και του κυρίου Ντεμαρνιακ και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορώ να είμαι τόσο ευγενής όσο ήταν οι συναδελφοί μου. Γιατί κάνατε μια δήλωση καλών προθέσεων ότι όλοι, αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο καθένας ήσασταν πάρα πολύ ασαφείς. Ούτε ένα αριθμητικό στοιχείο, ούτε μία λεπτομέρεια, ούτε ένα αποτεκτικό στοιχείο δεν μας δώσατε για το τι κάνετε, για το τι σκοπεύετε να κάνετε, για το ποια είναι τα πιο δυνατά σημεία και τα πια αδύναμα σημεία της στρατηγικής σας. Η κατάσταση στο Κωσικοπαίδιο και στη Βοσνία είναι δραματική. Ε, χρησιμοποιούμε και σπαταλούμε ε, χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν πήγατε χτες, πριν από δύο χρόνια πήγατε στην περιοχή. Δεν έχουμε λοιπόν βασικά στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε τον κύριο Μάρτι Δεν θέλουμε ο κύριος Μάρτι να ξέρει ποια είναι η κατάσταση. Η κατάσταση στο οργανωμένο έγκλημα στο Κωσυφοπέδιο είναι πιο παλιά και από τον πόλεμο στο Κωσυφοπέδιο. Είναι παλιό και γνωστό το πρόβλημα. Το ξέρουν και όσοι γνωρίζουν μόνο επιφανειακά την κατάσταση. Έχουμε εκεί από τις πιο δυνατές ε, οργανωμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Και αυτό το καταδεικνύουν όλοι, όλες οι έρευνες φαίνεται ότι το κοσυφοπέδιο αποτελεί κεντρικό σημείο όλων των οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Άρα, μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτά όλα τα αφήνετε κατά μέρο και μιλάτε για καλές προθέσεις μόνο και για ιδέες για το τι θα πρέπει να συμβεί στο μέλλον χωρίς να έχετε κάνει μια αξιολόγηση του παρελθόντο, χωρί να αξιολογήσετε αυτά που ήδη γνωρίζετε για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα στο Κωσυφοπέδιο. Να σας ερωτήσω λοιπόν, καταρχάς υπάρχει σαφέστατα ένα μεγάλο πρόβλημα ατιμορρησίας. Όλοι οι εισαγγελείς στο Κωσυφοπέδιο και έχω γνωρίσει αρκετούς, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να ερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και πολιτικής στο Κωσυφοπέδιο και πρέπει να γνωρίζουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία γιατί υπάρχει μεγάλο πλήθος στην κυβέρνηση του Κωσυφοπέδιου υπάρχει μεγάλη πίεση που ασκείται στον Πρωθυπουργό του Κωσυφοπεδίου ακριβώς λόγω εικαζόμενων σχέσεων με το οργανωμένο έγκλημα. Και θα πρέπει, θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι κάνει η Γιούλεξ προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την προστασία των μαρτύρων και μου προκαλεί μεγάλη μεγάλο αποτροπιασμό. Το κοσυφοπέδιο που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα δράσει. Ίσως και να κάνω λάθος, αλλά γι' αυτό είστε εδώ πέρα για να τα διευκρινίσετε αυτά, γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία με πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Αποτελεσματικό, το οποίο αποτελεί πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον μετά την ε, ε, διάσκεψη του Παλέρμο για το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Όλα αυτά λοιπόν ενισχύουν την κακή εικόνα που επικρατεί για τη χώρα και όπως ξέρετε υπάρχει και αυτό το σύστημα της ε, ε, περιτροπής του προσωπικού. Ξέρετε, αυτό είναι διοικητικό θέμα. Γιατί επιτρέπουμε στο θέμα αυτό, το είδα στο Κωσυποπέδιο πριν από 7 χρόνια ήδη. Γιατί δεν έχει αφαιρεθεί λοιπόν αυτή η διοικητική δυσκολία, αυτή η διοικητική απόφαση. Ποιο είναι υπεύθυνο εδώ στι Βρυξέλλε, είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε. Δεν μπορεί ο κόσμο να κάτσει να κάνει σοβαρή έρευνα σε έξι μόνο μήνε. Δεν είμαστε σοβαροί. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το παραμερίσουμε ω εμπόδιο. Και ύστερα έχουμε και το θέμα τη προστασία της εμπιστευτικότητα του απορρίτου. Δεν χρειαζόμαστε... Δεν χρειάζεται ο κύριος Μάρτιν να του πούμε ότι αν δεν υπάρχει προστασία του απόρριτου στο δικαστικό σύστημα δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Χάνονται μάρτυρες, δολοφονούνται μάρτυρες, ε, εκτοξεύονται απειλές κατά των, ε, των μαρτύρων. Γνωρίζουν όμως το κόσυφοπέδιο να πάσα στιγμή τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Εμείς πάλι με τη σειρά μας πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας σοβαρά δεδομένα και θα πρέπει να έχουμε και σοβαρά σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Κυρίλοφ, τελευταίος. Thank you, Chairman. Well, uh, I just uh, would like to continue. Am I right in understanding that... Μα συνεχίσω κι εγώ. Η αποκαλύψη του κύριου Μάρτη μας εξέπληξαν και τώρα ξαφνικά άρχισε να δουλεύει η αποστολή και ασχολείται για πρώτη φορά δηλαδή με το πρόβλημα της προστασίας των μαρτύρων. Διστάζω λιγάκι εδώ. Θα να ακούσω περισσότερα. Η βάση όλων αυτών είναι ότι έγινε πολύ νωρίς η αναγνώριση του κοσφοπεδίου. Και έτσι έδωσε τρομερές δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών ηγετών που στο παρελθόν ήταν αυτοί που έκαναν τον πόλεμο ε, στο κοσμοπέδιο και του οργανωμένου εγκλήματος. Τρομερές επαφές και συνδέσεις. Τώρα λοιπόν είναι στην κυβέρνηση αυτή η πολιτική και επομένως θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστορία, όχι μόνο για το κοσφοπέδιο. Νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν εκεί μολύνουν όλη την περιοχή. Αφορά αυτή η ιστορία όλες τις βαλκανικές χώρες. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Ακόμα και μια μικρή πρόοδος στο κοσφοπέδιο θα έχει θετική επιρροή και στις όμορες χώρες. Αλλά δεν υπάρχει πρόοδος. Αντίθετα, τα πράγματα επιδεινώνονται. Κάποια στιγμή θα υπάρχει κραγή κατάσταση. Και μετά θα ξυπνήσουμε και θα πούμε «Α, τώρα πρέπει να ανασκουμποθούμε». Και οι ηγέτε, όταν εμεί αποφασίσουμε να δουλέψουμε, θα πούνε Εσεί τι κάνετε εδώ πέρα, είμαστε ανεξάρτητη χώρα. Υπάρχουν τέτοια σημάδια. Για αυτούς τους τρεις, τέσσερις πράκτορες, τους Γερμανούς. Ξέρετε πολύ καλά πώς αντέδρασαν οι αρχές, η επίσημη ηγεσία σε αυτά που κάνανε. Πραγματικά ανησυχώ. Γιατί αν δεν υπάρξει πρόοδος σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το τομέα, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Υπάρχουν ήδη παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη ξέρετε για το γιο του πρώην Προέδρου. Έπειτα για το θέμα της προστασίας των μαρτύρων. Γίνεται να προστατεύσουμε τους μάρτυρες μέσα στο κοσφοπέδιο. Θέλω μια απάντηση. Και πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλόπενχάουρ και ο κύριος Ντεμαγνιάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση για την αφαίρεση των αρκών. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Για το γενικότερο, γενικότερη ανησυχία που εκφράστηκε, για ό,τι κάνει η Γιούλεξ για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι, είναι ότι θέλω να τονίσω ότι γίνεται σοβαρή η δουλειά από τη Γιούλεξ για να πολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Αν ενημερωθείτε, θα δείτε από, τα, από κόμματα του τύπου, από τις εκθέσεις του τύπου, ότι κάθε φορά που γίνεται μια ε, έρευνα ε, σε ένα σπίτι γίνονται συλλήψεις με σκοπό τη περαιτέρω έρευνας και διώξη. Το Δεκέμβριο του 2008 ε, ξεκινήσαμε να έχουμε κάποια επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ενώ τον Απρίλιο του 2009 είχαμε, φτάσαμε σε πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα, σε πλήρες επιχειρησιακό δυναμικό. Αν δείτε τον αριθμό των περιπτώσεων που η Ulex ε, διεκπαιρέωσε και υποθέσεις που ανέλαβε από την UNMIC, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Ε, μιλάμε για περιπτώσεις που έχουμε ερευνήσει, για υποθέσεις που έχουμε ερευνήσει. Υπάρχει μια συνείδηση τώρα στο κοσφοπέδιο ότι δεν υπάρχει πλέον τιμωρησία, γιατί πραγματικά δραστηριοποιείται η Γιούλεξ. Ακόμα και πολύ σημαντικές υποθέσεις που ερευνά η Γιούλεξ, τις προχωράει, υπάρχει πρόοδος. Φυσικά όλοι θα θέλαμε να κινούνται τα πράγματα πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχει μια αρχή που πρέπει να τη σεβόμαστε και τη σεβόμαστε πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Θέλουμε φυσικά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προστατεύσουμε την ε, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να αποφύγουμε πολιτικές παρεμβολές από πουδήποτε και προέρχονται. Αλλιώς οι έρευνε αυτέ θα γίνουν τελικά ένα πολιτικό παίγνιο στα πλαίσια τη ε, δικαστική διαδικασία. Και αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Αλλά ο επικεφαλή τη αποστολή θα σα ενημερώσει σίγουρα με περισσότερε λεπτομέρειε για τη δουλειά που γίνεται για το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά εμεί δεν αρκούμεθα απλώ σε δηλώσει ε, προθέσεων. Υπάρχει πραγματική πρόοδο. Για την προστασία των μαρτύρων τώρα. Το πρόγραμμα που έχουμε σε επίπεδο ULEPS είναι στεναρό αλλά δεδομένων των μικρών πόρων που έχουμε, έχουμε περιορισμένο δυναμικό εξορισμού. Ε, και αυτό εξαρτάται βεβαίως από την θέληση της χώρας να δεχτεί ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης μαρτύρων. Δηλαδή από την θέληση του κοσμοπεδίου να το δεχτεί αυτό. Θα σταματήσω εγώ εδώ και ο Ξαβιέ θα συνεχίσει. Ευχαριστώ. για το θέμα της προστασίας των μαρτύρων που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο από τον Νοέμβριο ήδη είχα συζητήσει πριν και από την έκδοση της έκθεσης του κυρίου Μάρτη, διότι φτάνοντας επικεφαλής αποστολής είδα ότι η κατάσταση δεν ήταν ιδεώδης ακόμη και παρά το γεγονό που όπω είπε ο Κέις έχουμε πάρα πολύ καλό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων που διαχειρίζονται εξαιρετικοί επαγγελματίες που έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη, αλλά έχει πρόβλημα προσωπικού. Δηλαδή, το πρόγραμμα αυτό και η ομβέλειά του που είχαν καθοριστεί από τα επιχειρησιακά ε, δράσεις που είχαν θεσπίσει στα κράτη-μέλη μειώθηκε αν θέλετε όσον αφορά την διάσταση του δεδομένου ότι πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο απαιτεί πολλούς πόρους, οι οποίοι λείπουν. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεχθούμε ευθύ εξ αρχής ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες. Πράγμα που καθιστά πρωταρχική σημασίας το relocation πρόγραμμα, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, μετακίνησης των μαρτύρων εκτός κοσυφοπεδίου, στο εξωτερικό. Δηλαδή, την βούληση των κρατών μελών να δεχθούν στην επικράτειά τους όχι μόνον μάρτυρες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις και την οικογένεια των μαρτύρων για απεριόριστη χρονική διάρκεια. Μπορεί να είναι καθόλου όλη τη διάρκεια της ζωής του ίδιου του μάρτυρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ λεπτό θέμα και κατανοώ ότι πολλές φορές κάποια κράτη-μέλη μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την αποδοχή αυτής της ε, έννοια της relocation και κυρίως πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους κυρίους, τους μάρτυρες, δεν είναι και παπαδάκια της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα και αν και μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό το relocation program. Όταν λοιπόν μου είπατε τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να μας συνδράμει, σας απαντώ το εξής. Επιμείνετε στις αρχές των κρατών μελών σας ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουν να δεχθούν στην επικράτειά τους αυτούς τους μάρτυρες. Βεβαίως δεν θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι θα υπάρχει και καμία πληθώρα μαρτύρων. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ε, για τι αριθμό μιλάμε. Κάποιος μάρτυρες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, δεν ξέρω πόσο ακριβώ, Πρόκειται όμω για ένα πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό θέμα και σήμερα πρέπει να πω ότι η δική μας αποστολή εξασφαλίζει με ικανοποιητικού όρου την προστασία των μαρτύρων, αλλά πρέπει να πω ότι έχει φτάσει και στα όρια τη όσον αφορά το θέμα τη δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα ε, της Όσον αφορά την ε, τοπική νομοθεσία του κοσυφοπεδίου. Όντω σήμερα Είμαστε ακόμη στο σχέδιο νόμου για την προστασία των μαρτύρων. Κατά την διάρκεια της πολιτικής αβεβαιότητας την οποία όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή την χρονική περίοδο κατά την οποία εγώ ήμουν επικεφαλής της αποστολής, το θέμα αυτό αποτέλεσε θέμα προτεραιότητος, χωρίς να γίνει τίποτα. Σήμερα επίσης είναι προτεραιότητα, θα το θέσουμε στην Δικαιοσύνης, αλλά πρέπει να σας πω ότι εκ του μηδενός η δημιουργία μιας υπηρεσίας αξιόπιστης προστασίας των μαρτύρων στο κοσυφοπαίδιο και το λέγω αυτό από την επαγγελματική μου πείρα θα χρειαστεί δύο με τρία χρόνια για να εφαρμοστεί. Και όποιος σας λέγει ότι χρειάζεται ο λιγότερος χρόνος δεν γνωρίζει την κατάσταση. Και αυτό είναι ένας από τους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε στο κοσυφοπέδιο, δημιουργήσουμε κίνητρα για να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι και τα δύο-τρία επόμενα χρόνια είναι προφανές ότι η διεθνής κοινότητα μέσω της αποστολής και ενός προγράμματος επανεγκατάσταση σε άλλες χώρες των μαρτύρων θα μπορέσουν από κοινού να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ τον Ξαβιέ. Τώρα όσον αφορά το προσωπικό. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας παράσχουν το προσωπικό που θα έχει τις γνώσεις να διεξάγει αυτές τις έρευνες. Βεβαίως έχουμε πολύ λίγους πόρους στη διάθεσή μας και από δικαστικής πλευράς. Ήδη 30% των ατόμων που χρειάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης έχουν αρχίσει να προσλαμβάνονται και θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό. Να επιτρέψουμε δηλαδή στα κράτη-μέλη να ε, προσλαμβάνουν προσωπικό εξειδικευμένο στον τομέα αυτό που το χρειαζόμαστε και όσον αφορά Uh, first of all, of course, uh, the tour of duty of Eulex personnel is not six months like in the military, but it's one year. Uh, but particularly in the prosecution side, even one year. Επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνιμο το προσωπικό. Καταρχάς προβλέπεται ένας χρόνος. Προσπαθούμε να παρατείνουμε την ε, παραμονή τους και πολλές ε, φορές υπάρχουν επικαλύψεις με κάποια σύμβαση μπορεί και να κρατήσει κάποιον και περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα επίσης να πω και να επιμείνω ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη και την άδεια των ε, κρατών μελών για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η Ρέλεξ ξέρουμε ότι θα πρέπει κάθε φορά να μας εξουσιοδοτεί να κάνουμε τις συμβάσεις που θέλουμε, να προσλαμβάνουμε προσωπικό, δεν είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι, μπορούμε να τα κάνουμε όλα από μόνοι μας, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε και θα πρέπει να ασκούμε πίεση για να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι, γιατί ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο για όλους εσάς. Θα ήθελα να επανέλθω στην έκθεση Μάρτη και στον τρόπο με τον οποίο τέθηκε σε κίνηση η αποστολή για να λάβει υπόψη το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την έγκριση και έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης έκθεση Μάρτη. Το ερώτημα που μου έθεσαν ευθύ εξ αρχή, επειδή είμαι υπεύθυνο αποστολή, είναι τι θα πρέπει να κάνει αυτή η αποστολή. Πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με την έκθεση αυτή, δεδομένου ότι αρχικά δεν υπάρχει καμία ορατή δεν υπήρχε καμία ορατότητα όσον αφορά τις ε, προθέσεις και των μεν και των δε. Ήταν λοιπόν η προσέγγιση μας μόνο δικαστική αν θέλετε και έτσι οι εισαγγελείς ασχολήθηκαν με το φάκελο αυτό όπως κάνουν συνήθως οι εισαγγελείς όταν κρίνουν ότι έχουν αρκετά στοιχεία, αρκετές μαρτυρίες ή αν υπάρχουν αιτιάσεις και ισχυρισμοί όπως αυτές της έκθεσης ε, Μάρτη που να αιτιολογούν κάτι τέτοιο. Από την δημοσίευση λοιπόν της έκθεσης Μάρτη πρέπει να πω ότι εγώ απευθύνθηκα στον κύριο Μάρτη όπως και η Εισαγγελής και άρχισε αυτή η προδικαστική έρευνα που όπως γνωρίζετε είναι κάτι το γενικό. Δεν στοχεύει σε κάποιον συγκεκριμένα, αλλά με γενικό τρόπο ε, μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος επιλαμβάνεται μίας υπόθεσης. Εγώ παρακολουθώ τους σύνεγγες στην όλη κατάσταση. Ξέρουμε ότι θα τη συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να χειριστούμε το θέμα αυτό. Εγώ ως επικεφαλής της αποστολής πρέπει να σας πω ότι δεν έχω να εκφράσω άποψη. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και είπαμε με τους εισαγγελείς ότι θα πρέπει να δούμε πώς προχωρεί η όλη αυτή ε, κατάσταση και πώς θα εμπλακούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Είπαμε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι ερευνητές και οι εισαγγελείς οι οποίοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ το θέμα αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς ασχολούνται και με άλλες τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις. Αλλά βασικά οι εισαγγελείς θα αφιερωθούν μόνο στην ε, έκθεση Μάρτη. Σιγά σιγά θα διευρυθεί όπως είπαμε ε, ο αριθμός των ε, εισαγγελέων και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε εκτός από τους κανονικούς ε, εισαγγελείς να προσλάβουμε και ίσως δύο-τρεις ε, περαιτέρω εισαγγελείς, πέντε-έξι εξειδικευμένους ερευνητές και κάποιους ε, δικαστικού βοηθούς για να μπορέσουν μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί εξ αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, αποφασίσαμε τα άτομα τα οποία θα επιληφθούν της υπόθεσης αυτής για λόγους ασφαλείας να ασχολούνται μόνο με αυτή την υπόθεση, να μην βρίσκονται στην, στα δικαστήρια στα οποία εδρεύουν κυρίως στην Αλβανία κάπου αλλού, να δημιουργήσουμε δηλαδή μια ειδική δομή ασφαλή και από ηλεκτρονικής πλευράς για να τους διασφαλίσουμε συνθήκες ασφαλείας άριστες. Και βεβαίως εκ παραλίλου τέθηκε ευθύς εξ αρχής το θέμα της προστασίας των μαρτύρων όπως προανέφερα έγιναν συζητήσεις πολύ θετικές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως για να εξασφαλίσουμε ότι την κατάλληλη στιγμή θα έχουμε και την ε, χρηματοδότηση που χρειάζεται για να προστατευθούν οι μάρτυρες αυτοί και κυρίως να μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να μετεγκατασταθούν, διότι όπως σας είπα χρονίζουν αυτές οι υποθέσεις, πρέπει να μεταγκατασταθεί και η οικογένεια και θα πρέπει να τους προσφέρουμε την ηλική υποστήριξη που χρειάζεται, πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Και πολλές φορές είπαμε χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν τέτοιου είδους υποθέσεις. Επίσης ήρθαμε σε επαφή με τις γειτονικές χώρες του Κωσυφοπεδίου που όπως γνωρίζετε φορώνται άμεσα από αυτή την υπόθεση και ιδιαίτερα στην Αλβανία, όπως ανέφερε και προηγουμένως η κυρία Πακ, που απήντησε λέγοντας ότι θέλει να συνεργαστεί ευχαρίστως. Έχω επιστολή του υπέξ της Αλβανίας που μας λέει ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί η Αλβανία και οι εισαγγελείς μας ήρθαν σε επαφή με τον ε, Γενικό Εισαγγελέα της Αλβανίας και όπως σας είπα είναι ενθαρρυντικές όλες αυτές οι επαφές και αποτελούν την βάση περαιτέρω ενεργειών μας στον τομέα αυτό. Στο θέμα τώρα της δικαιοδοσίας. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο, όχι μόνο εσά εδώ, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι όμως τα πράγματα αρκετά σαφή. Εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, ειδικό, ούτε Αλλά Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει έρευνες από μέρους της αποστολή στην Αλβανία. Την προηγούμενη Δευτέρα στην Πρίστινα άρχισε μία δίκη για κάποια ηγετικά στελέχη για κακομεταχείριση ε, από το 89 ε, κάποιων ατόμων που βρίσκονταν σε κάποια ε, ειδικά στρατόπεδα. Έχουμε εμείς τη δικαιοδοσία, έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο και κανένας δεν είναι αντίθετος στα πλαίσια της έκθεσης και της έρευνας θα κάνουμε μετά την έκθεση Μάρτη να κάνουμε και τέτοιου είδους έρευνες. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τους εξειδικευμένους Σέρβους εισαγγελείς εγκλήματα πολέμου, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα ή δυσκολίες και πρέπει να σας πω ότι οι δικοί μας εισαγγελείς με αυτούς τους εισαγγελείς ευθύς ε, εξ αρχής έχουν ε, τακτές επαφές για θέματα αγνοουμένων Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν έχουμε αρχίσει να ξεκαθαρίζουμε το γενικότερο τοπίο, ώστε να μπορούν οι εισαγγελείς μας να συνεργαστούν την κατάλληλη στιγμή και πρέπει να πω ότι ήδη έχουν υποβληθεί και κάποια αιτήματα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, εάν χρειαστεί να ξεπεράσουμε και την γεωγραφική επικράτεια αυτών των χωρών, και εδώ έχουμε τις κατάλληλες διαδικασίες, και οι εισαγγελείς μας έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν τέτοιου είδους διαδικασίες, πράγμα που σημαίνει ότι βεβαίως θα υπάρχει και βούληση και θετική συνεργασία εκ μέρου των αφορομένων και διαφερομένων κρατών. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι από δικαστική πλευράς είναι απόλυτα σαφής οι δικαστικές αρχές και εισαγγελεί. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόσκομα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που μπορείτε να έχετε για την έκθεση Μάρτη. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλές άλλες αναπάντητες. Εγώ προσπάθησα όμως να σας δώσω μια γενικότερη ιδέα του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την κατάσταση. Βεβαίως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις του θέματος εάν ληφθούν αποφάσεις στο α ή β επίπεδο που θα μας οδηγήσουν στο να αλλάξουν κάποια ε, θέματα σε αυτή την υπόθεση, τη στιγμή αυτή θα δουν πώς έχει προχωρήσει η προδικαστική έρευνα και σε ποιον θα πρέπει να την αποστείλουν οι δικοί μας Αλλά προς το παρόν έχει συμφωνηθεί κυρίως από τα κράτη-μέλη, τα οποία συνάντησα εγώ σε αρχές αυτού του μήνα στις Βιξέλλες ότι έχουν γίνει αποδεκτά αυτά τα οποία λέγουμε και συνεχίζουμε μέχρι να μας πει κάποιος «Στοπ, σταματήστε», εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση τόσο αναφορά τους αγνοουμένους που ανέφερε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Όντως, αγνοούνται ίσως περισσότερα από 1.800 άτομα, 1.821, για να σας δώσω και έναν ακριβή αριθμό. 1.821 άτομα, που όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, εξή, 1.400 Αλβανοί και 400 Σέρβοι περίπου. Δουλεύουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρσι πρέπει να πω ότι μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε γύρω στα 100 πτώματα τα οποία αποστήλαμε στις οικογένειές τους. Αυτό είναι δύσκολο μας. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε τις ε, κατάλληλες πληροφορίες για να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να μπορούμε εκ των υστέρων να κάνουμε ταυτοποιήσεις που μετά από 10 χρόνια από τα γεγονότα είναι πολύπλοκες. Αυτά γίνονται στο Department of Foreign Medicine με τη χρησιμοποίηση πάρα πολύ ε, πολύπλοκων αναλύσεων, DNA όπως γνωρίζετε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την κάθε οικογένεια και τι σημαίνει αυτό για την ε, περαιτέρω συμφιλή των διαφόρων εθνοτήτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 10 χρόνια μετά τα γεγονότα τα πράγματα είναι όλο και πιο πολύπλοκα, δεδομένου ότι ο χρόνος ενήργησε και πρέπει να σας πω ότι εδώ και 10 χρόνια κάναμε τα πιο απλά πράγματα με τον καλύτερο ή λιγότερο καλύτερο τρόπο. Σήμερα όμως πρέπει να χειριστούμε τις πιο δύσκολες υποθέσεις και η ταυτοποίηση των ατόμων που αγνοούνταν και βρέθηκαν είναι από τα πιο πολύπλοκα. Επίσης πρέπει να δούμε τι ε, συμβαίνει και με τις κλιματολογικές ε, συνθήκες που δεν μας βοηθούν. Σταματούμε το φθινόπωρο και ξαναρχίζουμε την ε, άνοιξη διότι καταλαβαίνετε ότι οι καιρικέ συνθήκες το χειμώνα δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να ενεργούμε Πρέπει όμως να αποδεχθούμε ότι τα πράγματα είναι όλο και πιο πολύπλοκα, αλλά κάθε χρόνο ε, ταυτοποιούμε όλο και περισσότερα πτώματα τα οποία έχουν ταφεί σε ε, μαζικούς κοινού τάφους και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το πολύ δύσκολο αλλά πολύ λεπτό και για τις οικογένειες. Ευχαριστώ. Δύο λόγια για τον Βορρά και το διάλογο. Καταρχάς για το διάλογο. Είναι μια ιστορική ευκαιρία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί η πολιτική πτυχή δεν είναι δική μου ευθύνη. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν την πολιτική σημασία και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει. Φυσικά, η διαδικασία θα είναι λεπτή. Ο διάλογος είναι σημαντικός και για το έργο της Γιούγκλαξ, γιατί μπορεί να βοηθήσει για να αφαιρεθούν κάποια εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα και παρεμποδίζουν το έργο μας ειδικά στο Βορρά. Έχουμε κάποιες ε, πρόοδους τώρα στα Μητρώα των ε, Πολιτών. Χρειάζεται να γίνει ως πρώτο βήμα διάλογος και ελπίζω ο διάλογος αυτός θα μπορέσει να θέσει και θέματα, να ρυθμίσει και θέματα τα οποία τώρα μας παρεμποδίζουν. Για το Βορρά, μας ρωτήσατε υπάρχει επιτυχία. Το θέμα είναι πώς τη μετράς την επιτυχία. Μία επιτυχία είναι ότι μέχρι στιγμής η Γιούλεξ κατάφερε να διατηρήσει τη σταθερότητα και συγχαίρω τη Γιούλεξ για την ε, καλή δουλειά και την K4 για την ε, καλή δουλειά που έκανε. Όπως είπε και ο Ξαβιέ, ο, επικε... ο επικεφαλής, υπάρχει μια task force στην Μήτροβίτσα. Ο που ασχολείται με εγκλήματα που έχουν σημασία για τον κόσμο. Ε, η EULEX ε, δεν είναι στρατός κατοχής, είναι μια αποστολή για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε αυτό το αίσθημα σιγουριά στο δρόμο. Συνεισφέρουμε λοιπόν και στη δημιουργία αυτού του αισθήματο ασφάλεια ε, για το σερβικό πληθυσμό στο βορρά. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν εγκληματικέ δραστηριότητε εκεί. Η αποστολή ξεκίνησε να κάνει κάποιε δράσει και σε αυτόν τον τομέα. Ξαβιέ, θα ήθελα να πει δύο λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ο Βοράς από την αρχή ήταν μια ζώνη προτεραιότητας για μένα όταν ανέλησα την κατάσταση τη στιγμή δηλαδή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Να πω ξεκάθαρα ότι σε καμία περίπτωση, και ξέρω ότι υπάρχει ο κίνδυνο, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δαιμονοποιήσω το βορρά. Σε καμία περίπτωση. Είμαι πολύ προσεκτικός και θα έχετε προσέξει ακούγοντά με να μιλήσω για τις προσπάθειες της Γιούλεξ στο βορρά τις προσπάθειες αυτές τις βάζω στο γενικό πλαίσιο προσπαθειών για το κοσφοπέδιο συνολικά. Κατά προτεραιότητα θέλω να καταπολεμήσω αυτό το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιείται στο Βορρά και που είναι διεθνικό. Αποτελείται από διάφορες κοινότητες συχνά οι κοινότητε βρίσκονται σε μια λογική ας πούμε πολιτικής και διοικητικής αντιπαράθεση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις εγκληματικέ δραστηριότητες συνεννοούνται απόλυτα οι κοινότητε για να κάνουν χρυσές δουλειές. Προσπαθώ λοιπόν να πείσω ε, τον πληθυσμό και δεν είναι εύκολο καθόλου ότι η θέληση, ότι η Γιούλεξ έχει τη θέληση να δείξει δικαιοσύνη ε, απέναντι σε όλες τις κοινότητες. Να είναι ισορροπημένη. Ο πρώτος στόχος, γενικός στόχος, είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος, να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και να αποφύγουμε την άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Ήμουν εκεί την άνοιξη του 2008 ως διοικητής της K4, την προηγούμενη ιδιότητά μου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει βία την αντιπαράθεση. Είναι λοιπόν ένας στόχος που προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε και δεν είναι πάντα εύκολο. Και μόνο με την καθημερινή μας παρουσία στο βόρειο κόσμο υφοπαίδιο μπορούμε να καταφέρουμε να την αποφύγουμε αυτή την αντιπαράθεση. Δεν λέω ότι κερδίσαμε. Αλλά αν δεν είμαστε παρόντες δεν θα τα καταφέρουμε. Όταν έφτασα στο κοσφοπέδιο πριν από τέσσερις μήνες, ποια ήταν η ε, πραγματικότητα της αποστολής. Πέντε ώρα το απόγευμα όλα τα μέλη της αποστολής ξαναπερνούσαν στο νότο. Και περνούσαν εκεί τη νύχτα τους ε, για να ξαναφύγουν το πρωί. Με εξαίρεση αυτούς που ήταν σε υπηρεσία, ας πούμε γύρω από την Μητροβίτσα κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι πηγαίναν σπίτι τους. Το πρώτο πράγμα που θέλησα να κάνω είναι να αυξήσω την μόνιμη παρουσία εκεί. Ε, δίνοντας κίνητρα στα μέλη της αποστολής και παροτρύνοντά τα να εγκατασταθούν ε, σε σπίτια κατοίκων στο βόρειο Κοσφοπέδιο. Όταν έφτασα, ήταν τέσσερα τα άτομα τα οποία ζούσαν στη Μητροβίτσα, στο βορρά. Ε, βόρεια από το Ιμπάρ. Σήμερα είναι 12 αυτά άτομα. Ίσως σας φανεί μικρή η πρόοδος, αλλά υπάρχει μια πρόοδος. Μην ξεχνάμε ότι χρειάστηκε και μας πήρε κάποιο χρόνο να προσαρμόσουμε τους κανόνες ασφαλείας που μας, επιβάλλει, που μας επέβαλε τότε το Συμβούλιο και τώρα η Επιτροπή, η, συγγνώμη, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και που πρέπει να εφαρμόσουμε αυτούς τους, νόμ, τους κανόνες. Ε, τους προσαρμόσαμε όμως και πιστεύω ότι μέχρι την Άνοιξη θα έχουμε 20 άτομα εγκατεστημένα σε σπίτια κατοίκων του Βορρά. Και με αυτόν τον τρόπο θα ζουν την, τη ζωή που ζει ας πούμε ο ντόπιο πληθυσμός. Όσοι έχουν επαφέ με τον πληθυσμό ας πούμε, και όσοι ασχολούνται με την ασφάλεια, καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει αυτό. Τώρα, δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφελεί ούτε υπερβολικά αισιόδοξοι. Χρειαζόμαστε χρόνο. Για να υπάρξουν μέτρα εμπιστοσύνη χρειάζεται χρόνο. Και ξέρω από εμπειρία ότι μερικέ φορέ κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προ τα εμπρό και ένα, μια θριαλίδα, α πούμε, μα πάει πίσω. Προ το παρόν έτσι πάνε τα πράγματα. Επίσης, επανοργάνωσα την αποστολή και στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου υιοθετήσαμε μία μόνιμη δομή. Η Task Force της Μητροβίτσα είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν ε, τελωνιακοί δικαστές, εισαγγελείς δηλαδή, ανακριτές, επίσης τελωνιακοί ανακριτές και εισαγγελείς, ούτως ώστε να υπάρχει ένα συγχρονισμός στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η δουλειά αυτή δίνει αποτελέσματα. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε μια επιχείρηση το Φεβρουάριο χρειάστηκε να τα αναβάλουμε λόγω της ε, προεκλογικής εκστρατείας στο τέλος του χρόνου, ε, που έδωσε καλά αποτελέσματα. Ε, οργα καταλάβαμε λίγο την οργάνωση και τις δομές που υπάρχουν. Έχουν και άλλους στόχους ε, και για το βορρά και για τον νότο του ΙΜΠΑΡ. Εμπλέκουμε και την τοπική αστυνομία. Γιατί είναι το καλύτερο μέσο δράσης και αντίδρασης. Πρόσφατα έκανε μία επιχείρηση εναντίον των ε, λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Πραγματικά ήταν επιτυχία. Ε, και την υποστήριξε και ο πληθυσμό ε, που πραγματικά θέλει να γίνουν τέτοιε προσπάθειε γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο ε, εξηγιένεται η ασφάλεια στον Βορρά. Ε, ανέθεσα στον βοηθό μου το ρόλο του εκπροσώπου μου, ούτως ώστε να πιέζει όλους τους φορείς να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτές τις προσπάθειες και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα απτά. Για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς. Γιατί είναι ένα ερώτημα που θέσατε αυτό της διαφθοράς. Ιδίω ορισμένε περιπτώσεις που ξεπίδησαν πέρυσι, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είμαστε μια αποστολή για το κράτος δικαίου. Είμαστε εκεί για να εφαρμόσουμε και να παροτρύνουμε, αν θέλετε, τους Κωσοβάρους να εφαρμόσουν το κράτος δικαίου με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και καλές πρακτικές. Μεταξύ των ευχολογίων και του δικαίου που μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα υπάρχει διαφορά. Οι έρευνες είναι μακρόπνοες αλλά γίνονται με σοβαρό τρόπο και Υπάρχει μια υπόθεση που θα την ξέρετε αν παρακολουθήσατε την επικαιρότητα. Θα είδατε ότι συμπληρωματικές έρευνες έγιναν, ε, ψάξαμε σε σπίτια, ε, κατασχέσαμε υλικό. Για προφανείς λόγους εγώ δεν μιλάω για τις τρέχουσες ε, δικαστικές διαδικασίες, αλλά υπάρχουν πράγματα που εξελίσσονται πραγματικά. Και όταν κοιτάζω τι γίνεται στην Ευρώπη, παντού, ε, για κάποιες βαριές και δύσκολες υποθέσεις, θέλω να σας πω ότι ένα χρόνο μετά είμαστε σε μια κλασική διαδικασία εξέλιξης μιας υπόθεσης διαφθοράς υψηλού επίπεδου ε, που είναι αρκετά ευαίσθητη. Δεν έχει κλείσει υπόθεση, δεν θαύτηκε η υπόθεση, οι εισαγγελείς δουλεύουν, οι ανακριτές δουλεύουν και την ε, κατάλληλη στιγμή θα φτάσουμε στο δικαστήριο με στοιχεία συγκεκριμένα. Επίσης ε, ξεκίνησαν κάποιες δίκες, η δίκη Γκέιτσι, ε, εκεί μιλάμε για εγκλήματα πολέμου περισσότερο. Αλλά έχετε και την υπόθεση μεντικιούς που ακούστηκε πολύ ε, στον τύπο κτλ. Υπάρχουν υποθέσεις λοιπόν που φτάνουν στην δικαιοσύνη. Υπάρχουν υποθέσεις που ξεκίνησαν το 2010 που φτάνουν στα δικαστήρια σήμερα για να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης. Τώρα, τι αποφάσεις θα πάρουν οι δικαστές. Σας παραπέμπω στις στατιστικές ε, και στις καλές πρακτικές στην Ευρώπη. Ε, στην Ευρώπη όλες οι δίκες δεν καταλήγουν σε κατάδειξη, σε, κατα... <laughs> Συγγνώμη, σε καταδίκη. Υπάρχουν υπάρχουν και οι δικηγόροι κτλ. Το γεγονό ότι παραπέμπεται κάποιο ενώπιον του δικαστηρίου δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται οπωσδήποτε. Το ξέρετε όλοι. εμείς ένα τμήμα τη αποστολής μας, ας πούμε, ε, ένας λόγο που είμαστε εκεί είναι για να δώσουμε και το, καλό παράδειγμα στις ε, τοπικές αρχές. οι σχέσεις με την κυβέρνηση σας ταράζουν. Σε ποιον αναφέρεστε. Εκτός μικροφώνου, κυρία Πακ. Δεν ξέρω αν παλιοί υπάλληλοι της ΟΝΜΙΚ έχουν εμπλακεί στην πολιτική. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν πρώην ε, υπάλληλοι της ΟΝΜΙΚ που σήμερα ασχολούνται με τη δική μας. Ε, έχουν προσληφθεί δηλαδή από την Ulex. Αλλά κάποια στιγμή άνοιξε η αποστολή, μεγάλωσε και χρειάστηκε να προσλάβουμε και ανθρώπους ε, από την περιοχή, δηλαδή για τη μετάφραση, για διάφορους λόγους, εν Ο προκάτεχός μου ήταν πολύ προσεκτικός. Ήθελε η Γιούλεξ να ξεκινήσει μετά μπουλαράζα. Υπάρχει και ένας λόγος, ο τρόπος που μας αντιμετώπιζε εκείνη η κοινή γνώμη. Αλλά τελικά χρειάστηκε να μετριάσει αυτή την προσέγγιση, έτσι, την τρομερά ρήξη και και αναγκάστηκε ας πούμε να προσλάβει και προσωπικό, παλιό προσωπικό της UNMIC. Αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως επωφεληθήκαμε και από την εμπειρία ανθρώπων που γνωρίζανε κάποια πράγματα, που ήταν από εκεί κτλ. Τώρα, αν υπάρχουν πρώην υπάλληλοι τη UNMIC, οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική, δεν έχω ιδέα. Θα δω θα το κοιτάξω, θα το ψάξω και θα δω τι διαστάσεις έχει πάρει αυτό το φαινόμενο. Πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Αουλάκη, θέλετε πολύ συγκεκριμένη ερώτηση να κάνετε σύντομα, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Πρόεδρε, μία ερώτηση θα κάνω και μία σύντομη παρατηρήση. Γιατί ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση της Γιούλεξ. Θεωρώ ότι πραγματικά δεν οδεύεται πουθενά. Γιατί σας λείπει ε, το βασικό νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό δεν φταίτε εσείς. Ε, και δεν μπορείτε να καταπολεμήσετε το οργανωμένο έγκλημα και να φροντίσετε και την προστασία μαρτύρων. Αν δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι νόμοι, αν δεν υπάρχουν νόμοι για την προστασία μαρτύρων, όχι μόνο για να μπορέσουν να κρυφτούν τα άτομα αυτά, αλλά για να διασφαλιστεί ότι το κράτος δικαίου ισχύει και για αυτούς. Αν δεν, υπάρχουν, ε, αν δεν υπάρχει κατάργηση του απορρίτου των τραπεζών, αν δεν υπάρχει ε, των περιουσιακών στοιχείων, ξεκινήσαμε το 1996 είχαμε τη σύμβαση του Παλέρμο, το, η οποία διασφάλιζε ότι τηρούνται αυτές οι αρχές από όλα τα προσωπογράφοντα κράτη. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, πολύ απλά δεν θα μπορέσετε να καταφέρετε τίποτα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ούτε στο Κωσυφοπέδιο, ούτε πουθενά αλλού. Άρα, έχετε εισαγγελεί εκεί, οι οποίοι δεν σας προτείνουν μία στρατηγική σαφή και ακολουθείτε μία προσέγγιση έτσι επιφανειακή και είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη το θέμα αυτό. Και ασφαλώς υπάρχει και το θέμα των πόρων που δαπανάτε. Ερωτώ λοιπόν κύριε Κλόπενχάουερ, πόσο κόστησε, ποιος ήταν ο προϋπολογισμός της Γιούλεξ έως τώρα, στα δύο χρόνια πλήρους λειτουργικότητάς τους και ποιο Ποιο είναι ο προ... υπολογισμό που προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια, πόσα άτομα απασχολείτε και σε ποια θέση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να πω ότι η EULAX ε, είναι εκεί για να εφαρμόσει το δίκαιο που υφίσταται και συμφωνώ ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο. Δεν διαφωνώ καθόλου με τον κύριο Αρλάκη. Και αυτό ισχύει όχι μόνο στο Κοσμοπέδιο, αλλά και στη Βοσνία και σε άλλα μέρη για να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά η αποστολή μας είναι να εφαρμόσουμε το δίκαιο. Αυτό έχουμε ως εντολή για το κόστος. Ε, ε, εκτιμώ 150 εκατομμύρια ευρώ είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός, ίσως και κάτι παραπάνω. Και τώρα απασχολούμε μεταξύ ε, περίπου 700 άτομα. Οι πιο πολλοί είναι αστυνομικοί λόγω μεταξύ άλλων και των εκτελεστικών καθήκοντων της αποστολής. Αυτά είναι λοιπόν τα αριθμιστικά στοιχεία. Είναι όμως κατά προσέγγιση γιατί δεν έχω ακόμα λεπτομέρειες. Και πόσους εισαγγελείς, ρωτάει ο κύριος Αρλάκη. 27, 27. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η συζήτησή μας για το κοσυφοπέδιο. Σας ευχαριστούμε θέλουμε να ενημερωνόμαστε τακτά διαστήματα για τις δραστηριότητες των αποστολών σας. Θέλουμε λοιπόν να επαναλαμβάνουμε τέτοιου είδους ε, συναντήσεις μαζί σας και κυρίως αν υπάρξουν και θέματα προτεραιότητας. Σας ευχαριστούμε. Ε, ζητώ συγγνώμη, υπάρχει καθυστέρηση στο όλο πρόγραμμα, αλλά καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον το θέμα. Τώρα δίδω το λόγο στον κύριο Φέλλερ, κεφαλής αντιπροσωπείου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα. Αξιότιμοι βουλευτές. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου που έρχομαι εδώ να σας ε, ενημερώσω για την εξέλιξη της ε, αστυνομικής αποστολής και την, ε, τα επιτεύγματα που έχουμε σημειώσει σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η κατάσταση στη Βοσνία Ζεγοβίνη εξακολουθεί να είναι περίπλοκη, όπως ξέρετε, και με την στρατιωτική αποστολή μας έχουμε την ίδια εκτίμηση της κατάστασης ως προς την ασφάλεια παρά την παρατεταμένη, τα παρατεταμένα πολιτικά προβλήματα της μεταεκλογικής περίοδου και της οικονομικής κρίσης. Δεν υπάρχουν δείκτες που να υποδεικνύουν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση ως προς την ασφάλεια. Ωστόσο σημειώνουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη αίσθηση ανασφάλειας λόγω των εγκλημάτων κατά των περιουσιακών στοιχείων και λόγω της ιδιαίτερης ε, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης πολλών πολιτών. Για λεπτομέρειες ε, της αποστολής μας. Σας ενημέρωσα πέρσι το καλοκαίρι και σας ανέφερα ότι είχαμε πετύχει ένα ορόσημο τον Απρίλιο του 2008 το πακέτο μεταρρύθμισης που άνοιξε το δρόμο για την Συμφωνία ατερική Σχέσης. Η σχετική συμφωνία για την απελευθέρωση του καθεστώτος ε, θεωρήσεων και το 2010 και καταβάλαμε προσπάθειες για την κοινή οικοδόμηση ε, δυνάμεων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και τονίζω εδώ το κοινό γιατί να σας υπενθυμίσω ότι στη Βοσνία Ερσεγοβίνη υπάρχουν 17 υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου που εμπλέκονται. Έχουμε 80 λοιπόν ε, εμπειρογνώμονες ε, αστυνομικούς, 40 υπαλλήλους ε, δημόσιας διοίκησης και περίπου 150 επαγγελματίες και γενικό προσωπικό από τη Βοσνία Ριζεκοβίνη το 2010 ήταν σημαντικό έτος και πολύ επιτυχές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας η απόφαση του Συμβουλίου να αρθούν οι απαιτήσει για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντική. Το 2010 γνώρισε πολύ καλά οργανωμένες δράσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Διοργανώθηκαν και εκτελέστηκαν περισσότερες από 30 τέτοιες απόστολες κατά σημαντικών μορφών οργανωμένου ε, εγκλήματος και εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Τον προηγούμενο, μάλλον τον τελευταίο μήνα το 2010, από τον Οκτώβριο στον ε, Δεκέμβριο, έγιναν δύο πολύ σημαντικές δράσεις ε, κατά του οργανωμένου εγκλήματος και ε, συλλήφθησαν ε, αστυνομικοί και αξιωματούχοι υψηλού επίπεδου. Άρα, ποια είναι τα συμπεράσματα λοιπόν από, τα, από τις εξελίξεις αυτές. Καταρχάς, ότι οι αρχές έχουν τροποποιήσει το πλαίσιο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων λόγω και του οδικού χάρτη για τις θεωρήσεις και πλέον καταδεικνύουν την ικανότητά τους να πετυχαίνουν αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούν οι συζητήσεις στο πρόβλημα των ε, μηχανισμών λογοδοσίας και των αναγκών συστηματικής και συνολικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα το εξηγήσω και σε λίγο. Οι συλλήψεις του Δεκεμβρίου στο καντόνι της Ουνασάνα, η αποστολή Κάσλ, είχαν στόχο την ηγεσία της αστυνομίας και η αποστολή τάξα οδήγησε στη σύλληψη σημαντικού αριθμού πολιτι... Ε, αστυνομικών της ε, συνοριοφυλακής. Ε, χρειάστηκε να επιστρατεύσουμε την αποφασιστικότητα και της αστυνομίας και των εισαγγελέων για να μην μείνει κανείς ατιμόρυτος. Έχουν αρχίσει λοιπόν να πετυχαίνονται αποτελέσματα από τις κοινέ αυτές δράσεις και η συνεργασία μεταξύ εισαγγελέων και αστυνομίας μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά έχουν βελτιώσει την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η αποφασιστικότητα κυρίως ε, του Γενικού Εισαγγελέα θα πρέπει να επενεθεί. Γιατί συχνά συζητώ μαζί του και θα πρέπει πραγματικά να τονίσω την αποφασιστικότητά του. Αυτό τρία στοιχεία εξηγούν τα επιτεύγματά μας. Καταρχάς, ε, διάλογοι, ο διάλογος για τις θεωρήσεις βελτίωσε γενικότερα το συνολικό σύστημα. Κατά δεύτερον, η συνεργασία, κανονική συνεργασία των υψηλών αξιωματούχων απέδωσε πρώτους καρπούς σε περιπτώσεις, ε, για παράδειγμα, διαφθοράς, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν καταλήλως, γιατί τρίτον, η συνολική ικανότητα έχει αυξηθεί και αυτό είναι μια λογική απορία και των εγχώριων προσπαθειών, αλλά και των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας τα τελευταία δεκαετία. Άρα, κάπως προχωράμε, κάπως προχωράμε και πλησιάζουμε το στόχο μας. Ωστόσο, δεν αρκούν αυτά που έχουμε πετύχει ακόμα σε ό,τι αφορά και τις φιλοδοξίες της ε, Βοσνίας Ριζεγοβίνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το 2011 θα εργαστούμε κυρίως επί στρατηγικού και θεσμικού επίπεδου προκειμένου αυτές οι προσπάθειες να καταστούν βιώσιμες και οι δράσεις να καταστούν ε, να υπάρχει να είμαστε υπόλογοι. Καταρχάς λοιπόν σε περιφερειακό επίπεδο και κρατικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο καντονιών θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία. Η συνοριοφυλακή, οι αρχές έμεσης φορολογίας, τα τελωνία και όσοι είναι υπεύθυνοι για θέματα μετανάστευσης αποτελούν τα άτομα τα οποία θα πρέπει να εργαστούμε για την εφαρμογή των νομοθεσιών τα, οι πιο καινούργιες υπηρεσίες θα χρειαστούν τεχνική αρρωγή και πολιτική δέσμευση από τις ε, χώριες αρχές αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους εταίρους. Οι τακτικές ανεπίσημες συναντήσεις ε, της αστυνομίας και των εισαγγελέων συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να θεσμοθετηθούν και αυτή η ανάγκη για θεσμοθέτηση θα αποτελέσει ένα βασικό ζήτημα το, την επόμενη περίοδο και θα αποτελέσει και μια σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Σε υπουργικό επίπεδο, το Υπουργείο Ασφάλειας βελτιώνει την, το συντονισμό του κλάδου, ιδιαίτερα σε κλάδους που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που άπτονται και διεθνών συμβάσεων το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν να υπάρξουν ειδικοί μηχανισμοί εποπτείας για τις πέντε ε, χώρες των Βαλκανίων για τις οποίες και το καθεστώς ε, θεωρήσεων. Και αυτό θα διασφαλίσει μια βιωσιμότητα στις προσπάθειες αυτές και η διαϋπουργική, τα διαϋπουργικά στοιχεία θα πρέπει να ενισχυθούν. Αυτή είναι στρατηγική στόχη όταν θα σχηματιστούν κυβερνήσεις. Κατά δεύτερον, η λογοδοσία, ένα θέμα το οποίο επανέρχεται διαρκώς ε, στο επίκεντρο στην ασάνα η θεσμική διάσταση αναγνωρίζεται ότι επί σειρά ετών ε, συμμετείχαν υψηλοί αξιωματούχοι σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Ποια είναι λοιπόν τα μαθήματα τα οποία διδασκόμαστε από το παρελθόν. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέσουμε στις αρμόδιες κυβερνήσεις και στα αρμόδια κοινοβούλια. Η δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, προαπαιτεί και μια διαρκή, ένα διαρκή έλεγχο των διοικητικών ε, ρυθμίσεων και ενδελεχή εξέταση υποθέσεων απάτης, ε, διαφθοράς και φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να ρωτηθούμε γιατί δεν καταγγέλουν οι πολίτες τέτοιες περιπτώσεις διαφθοράς και θα πρέπει να εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο και τις ε, ελλείψεις τους αλλά βασικά θα πρέπει να αποσταλεί ένα έντονο μήνυμα από την εκτελεστική εξουσία προς τους πολίτες ότι οι πολίτες μπορούν να εμπιστεύονται και το UPM και την απόστολη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά και θα είναι μία από τις προτεραιότητές μου να διευκρινίσουμε ότι κοιτάξτε καλά όσα κάνετε αλλά θα πρέπει να υπάρχουν διαρκείς προσπάθειες. Η βιωσιμότητα και η λογοδοσία είναι τα κλειδιά για την επιτέξη της αποστολής μας και γι' αυτό μία αποστολή κράτους ένα σύστημα κράτους δικαίου το οποίο δεν είναι βιώσιμο θα παραμείνει κλώτσο σκούφι της εκάστοτε ε, κυβέρνησης και ένα σύστημα δι, ε, κράτους δικαίου το οποίο δεν είναι υπόλογο στους πολίτες ε, υπόκειται στον κίνδυνο της διαφθοράς. Θα πρέπει να είναι βιώσιμο και να υπάρχει λογοδοσία. Ιδάλλως όλοι θα προσπαθήσουν να το υπονομεύσουν. Δεν είναι περίεργο αυτό και η βασική αντίδραση στις προκλήσεις αυτές θα πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο γιατί ε, υπάρχουν βασικά πολιτικά είναι τα κριτήρια για τη διαδικασία προσχώρησης. Ωστόσο, η πολιτική διαδικασία και αυτή υποφελείται από τη λογοδεσία και την βιωσιμότητα. Και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αξίες για την προστασία του κράτους δικαίου. το εφιστάμενο πολιτικό σύστημα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μπορεί να σπάσει το σύστημα εφαρμογής του νόμου το οποίο επικρατεί και εμείς ε, προσπαθούμε από, διεθνής, ε, από διεθνούς άποψης να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα για να δώσει κίνητρα για την συνοχή προκειμένου να εξευρεθούν κοινέ λύσεις για να προσεγγίσει η χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αποστείλουμε ένα μήνυμα σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες μέσω μιας ισχυρής πολιτικής παρουσίας και εκ παραλίλου θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή μέσω στρατηγικών συμβουλών αλλά και μηχανισμών τεχνικής αρρωγής που είναι απαραίτητη στον τομέα της εφαρμογής της, ε, του νόμου και του δικαίου. Και τέλος, τέλος είμαι αισιόδοξο ότι η στρατηγική αναθεώρηση του Συμβουλίου θα παράγει έναν ισχυρό μηχανισμό πέρα από την εντολή του UPM που όπως ξέρετε θα λήξει στα τέλη του 2011. Εκ παραλλήλου, η αποστολή υποστηρίζει ήδη εισερχόμενες ομάδες ε, μέσων για IPAs, για χρηματοδοτούμενα τεχνικά προγράμματα. Ευχαριστώ λοιπόν Πρόεδρε για την προσοχή σας. Merci, ε, euh, Σε ευχαριστώ κυρία Πάκ. Κύριε Φέλλερ, ακούγοντας αυτά που μας λέτε θα μπορούσα σχεδόν να σας πιστέψω. Ωστόσο, νομίζω ότι η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Σας εύχομαι να ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζετε. Όμως ξέρετε σε ποιο περιβάλλον ζείτε, σε ποιο συνταγματικό περιβάλλον ζείτε. 17 αστυνομικέ υπηρεσίες, 13 ε, υπουργοί ε, Όλα πολλαπλασιάζονται και μιλώντας μόνο για το καντόνι του Νασάνα όπου κάτω αποκαλύφθηκε. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 9 καντόνια και υπάρχουν και άλλες οντότητε. Δεν μπορείτε να είσαστε πανταχού παρόν. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς θα τα καταφέρουμε στη χώρα αυτή πραγματικά να δημιουργήσουμε κράτος δικαίου όσο δεν υπάρχουν κοινές, ε, κοινοί θεσμοί οι οποίοι θα απολαμβάνουν το σεβασμό όλων. Πάντα θα αμφισβητούνται αυτοί οι θεσμοί. Πώς θέλετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά όταν τα μέτρα σας δεν γίνονται καν αποδεκτά. Και σας λένε ότι κοιτάξτε δεν σας αφορά το θέμα αυτό γιατί αυτό γίνεται στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό γίνεται και στη μία οντότητα αλλά και στην άλλη οντότητα. Στη μία οντότητα βγαίνει και λέει ο ένας ότι είναι αρμόδιος, αλλά στην άλλη βγαίνει ένας άλλος αρμόδιος και ε, φάσκουν και αντιφάσκουν. Αυτό πραγματικά είναι το μεγάλο πρόβλημα, το συνταγματικό που αντιμετωπίζετε και εσείς στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Πριν από ε, κάποια χρόνια υπήρξε η μεταρρύθμιση του αστυνομικού σώματος. Το είχαμε καταστρώσει αυτό το σχέδιο, πάρα πολύ όμορφο αλλά μια τέτοια αστυνομική μεταρρύθμιση όπως κάναμε τότε από τον πρώην συνάδελφο Μάρτιν για μια χώρα όπως η Βοσνία Ερζεγοβίνη για μια χώρα όπως η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ε, ωφέλιμο και θεωρώ ότι ήταν και αποτυχημένο και τελικά προέκυψε αυτό που είχαμε ότι αυτό που είχαμε απαιτήσει τότε ήταν πραγματικά γελίο. και τελικά μας οδήγησε στην αποδοχή της συμφώνου ε, με εταιρικής σχέσης. Αμφιβάλλω όμως ότι χωρίς θεσμικά όργανα ε, στη χώρα αυτή, ε, θεσμικά όργανα τα οποία απολαμβάνουν το σεβασμό όλων, μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε. Όση δουλειά και να κάνετε μέχρι το 2011 θα φύγετε από μια χώρα τελικά όπου θεωρώ ότι το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν θα έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα. Όχι επειδή εσείς φταίτε, φταίει η κατάσταση φρικτή με τα θεσμικά όργανα. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα κυβέρνηση. Γιατί οι πολιτικοί δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν για να ακολουθήσουν μια κοινή διαδικασία. Η διαδικασία προσχώρηση θα μπορούσε ενδεχομένω να βοηθήσει, αλλά έχω την εντύπωση, κοιτώντα και την πολιτική κατάσταση, ότι δεν του νοιάζει του πολιτικού. Και αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, ότι το θέμα δεν είναι να βοηθήσουν τον κόσμο, του νέου στη χώρα, να καταστήσουν πιο ελκυστικό το επενδυτικό περιβάλλον, για, με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ε, δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσείς δουλεύετε πολύ σκληρά, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ταμιευτεί η δουλειά σας και να επιτευχθούν είτε μεγάλες είτε μικρές αλλαγές. Πολύ απλά δεν έχουμε θεσμούς σωστούς. Ο ένας λέει το ένα, το άλλο λέει το άλλο. Ο ένας λέει αριστερά, ο άλλος λέει δεξιά. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και γι' αυτό πολύ λυπάμαι γιατί δουλεύετε πολύ σκληρά και με πολύ μεγάλη συμπάθεια στη χώρα αυτή. Αυτό όμως δεν ε, το, δεν το δέχεται η πολιτική κατά πραγματικότητα, παρόλο που ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά. Θα ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω, αλλά δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Κυρία Κοπά. Δυστυχώ, οι περισσότεροι συμφωνούμε με αυτά που τώρα μόλι είπε η κυρία Πακ. Δυστυχώ, δυστυχώ την χώρα. Και ευτυχώς εμείς συμφωνούμε. Το ερώτημά μου είναι διαφορετικό. Πώς αξιολογείται την συνεργασία της Βοσνίας Ερσεγαβίτης με τις γειτονικές χώρες. Υπάρχει κάποια αλλαγή τους πρόσφατους μήνες ή έχετε την ίδια κατάσταση με αυτή η οποία εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλισεν. Just being called from another committee meeting. <laughs> It's busy today. με πήραν από κάποια άλλη επιτροπή. Κι εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτό που είπε κυρία Πακ. Πολύ θετική φαίνεται η ιστορία σα, αλλά φαίνεται ότι έχετε μια επιτυχημένη αστυνομία ένα, σε μια χώρα που δεν λειτουργεί που δεν υπάρχει. Όσο προχωρούμε, τόσο χειρότερα είναι αυτά τα οποία ακούγονται και οι απειλές οι οποίες εκφράζονται. Οι προκλήσεις και κυρίως το γεγονός ότι τίποτε δεν δουλεύεις όπως θα έπρεπε σε ένα κράτος δικαίου. Με απασχολούν λοιπόν και περισσότερο αυτές οι καταστάσεις. Αποτυχημένο κράτος θα είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη κάποια στιγμή. Και πώς έχει σχέση με αυτά τα οποία αποκομίζουμε εμείς ως εντύπωση με αυτά τα οποία είπατε εσείς. Ο κύριος Σαλάκη. παρεμφερεί ερωτήματα με αυτά που έκανα για το κοσυφοπαίδιο. Παρεμφερεί τα πράγματα και εδώ. Παρά το γεγονός ότι εδώ ίσως είναι χειρότερα τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι ακούμε στους τίτλους των εφημερίδων για το κοσυφοπαίδιο. Πιστεύω, έχοντας σας ακούσει επίσης, ότι η αποστολή δική σας έχει τρομερές εξουσίες. Και την δύναμη να παρέμβει στις πολιτικές διαδικασίες και να χρησιμοποιήσει ισχυρά μέτρα. Ίσως αυτό να μην είναι πάντα πολύ θετικό, αλλά πολλές φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε κράτος δικαίου και ακόμη και αν υπάρχει πολλές φορές δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι καταπολέμησης διαφθοράς. Πείτε μου εσείς, για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε στη Βοσνία το οργανωμένο έγκλημα για τη διαφθορά, τι είδους μέσα χρησιμοποιείτε. Διότι ε, δεν το κατάλαβα. Μιλάμε για δύο χώρες που είναι στην Ευρώπη, που κάποιες από αυτές θέλουν να γίνουν και μέλη της Ευρώπης και έχουμε το εξή ε, παράδοξο. Ό,τι συνέβη στην Ευρώπη για το ξέπλυμα χρήματος, τα τρία τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, το ξέπλυμα χρήματος, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, φαίνεται ότι γίνεται εκτός Κωσυφοπεδίου και Βοσνίας. Δηλαδή έχουμε ευρωπαϊκές κανόνες και προδιαγραφές για να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε στις περισσότερες χώρες μέλη ισχυρά μέσα για να τα καταπολεμήσουμε και φαίνεται ότι εκεί δεν ισχύουν αυτοί οι κανόνες. Το ερώτημα μου, τα ερωτήματα μου λοιπόν είναι τα εξή. Ποια είναι η νομοθεσία για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, για την προστασία μαρτύρων, για τη ε, διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων. Και αν δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που αφορά τις ε, συνωμοσίε, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά. Επίσης, ποια είναι η δύναμη που έχουν οι δικαστικές και οι εισαγγελικέ αρχές για την κατάσχεση των ε, περιουσιακών στοιχείων των διεφθαρμένων ατόμων. Υπάρχουν λοιπόν σε όλο τον κόσμο, την Δυτική Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά τον κόσμο, ισχυρά μέσα που διαθέτουμε για να καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά. Και τι γίνεται, κάνουμε κουβέντα, μπλα μπλα μπλα, όπως ο τύπος αναφέρει, πολιτική διαφθορά και δεν ξέρουμε τίποτα σε ποια κλίμακα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ποια είναι τα ποσά τα οποία θα μπορούσαμε να επενδύσουμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά. Τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγέ. Δεν θέλω να σας επικρίνω πολύ, αλλά σας παρακαλώ να είστε πιο συγκεκριμένο και να μας πείτε πώς αξιολογείτε βάσει αυτών που σα είπα την κατάσταση στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ευχαριστώ. Έχουμε 10 λεπτά για να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις και όπως διευκρίνησαν και κάποια μέλη, υπήρξαν και σχόλια, δεν χρειάζεται να απαντήσετε, αλλά τέθηκαν και ερωτήσεις και σας ευχαριστώ που θα απαντήσετε. Κύριε Κλάπενχάουερ, θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Είναι πολύ πλούσια αυτή η συζήτηση. Δέχομαι τις επικρίσεις και θετικά. Διότι πραγματικά από πολιτικής πλευράς δεν υπάρχει πρόεδρος, από νομοθετικής ναι. Εμείς πρέπει να πω ότι έχουμε να κάνουμε και με τεχνική, συμβουλευτική απόστολη. Και σωστά λέτε ότι θα πρέπει να δούμε σε ποια πλαίσια κινούνται οι αποστολές των οποίων ηγούμεθα. Όντως θα πρέπει να βελτιθούν πολλά πράγματα. Συμφωνώ κι εγώ, δεν διαφωνώ. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ ανάλυσης κατάσταση μεταξύ του τι μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι η εντολή μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δώσω στο Στέφαν το λόγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έγιναν συγκεκριμένα. Σα ευχαριστώ, κυρία Βουλευτή, για τις ερωτήσεις σας. Θα κάνω το πρώτο σχόλιο μου στα γερμανικά. Δεν μπορώ να αντιτάξω τίποτε στα επιχειρήματά σας. Μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει αντίθετη σύνταξη της δικής αξιολόγησης και των δικών μας λεγόμενων. Όντως, είμαστε μια τεχνική αποστολή που ενεργεί μέσα σε ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό γενικότερο κλίμα. Αυτό είναι αληθές. Άρα θα πρέπει να λαμβηθεί υπόψη αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα για να απαντήσω. Και αν μου δώσει 10 λεπτά ο πρόεδρος, δηλαδή μου διπλασιάσει το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα μπορούσα να σας μιλήσω για αυτά τα θέματα πιο λεπτομεριακά. Σας ε, μίλησα προηγουμένως για την περιοχή του Σάνα. Δεν θα πρέπει, δεν, θέλω, δεν αναφέρθηκα σε λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να πω ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθούμε με ενδυμικά προβλήματα ή με προβλήματα που αφορούν τα διαφορετικά καντών, διαφορετικές περιοχές γενικότερα. Και μετά από τα σχόλια που έγιναν, θα πρέπει να πω ότι δεν πρέπει κανένας να πλήσεται από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και γίνουν εκεί. Για τη διαφθορά, για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, Πώς ενεργούμε. Εντοπίζουμε το πρόβλημα και παρεμβαίνουμε σχολιάζοντας για να δούμε αν από ψυχολογικής πλευράς μπορούμε να, κάνουμε, να έχουμε κάποια αλλαγή και βλέπουμε πώς έχει το πρόβλημα. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενεργήσουμε. Ποια είναι τα πιο κατάλληλα μέσα που διαθέτουμε. Έχουμε, όπως σας είπα, μέσα στη διάθεσή μας, αλλά εμείς έχουμε συμβουλευτικό τεχνικό ρόλο. Και σε επίπεδο αστυνομίας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αν θέλετε. Στο κοσυφοπέδιο ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ξέρουμε ότι το συντομότερο δυνατό έπρεπε όλες οι εξουσίες δικαιοδοσίες να περάσουν σε τοπικό επίπεδο. Αλλά σας λέγω ότι η δική μας η προσέγγιση είναι τεχνική. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Πήγα στην Πανιαλούκο, πήγα στην Τούσλα, θα πάω και σε άλλες χώρες για να μιλήσω με τους επικεφαλείς των αστυνομιών για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν πρέπει επίσης να πιστεύετε ότι όλα είναι η άσπρα ή μαύρα στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Υπάρχουν πολλοί τόνοι του γκρι και πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν για να προχωρήσουν τα πράγματα. Πρέπει επίσης να σας πω ότι το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο τόσα χρόνια μετά από το τέλος των δημαχών. Και δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να προχωρήσουμε, να ενεργούμε συντονισμένα, να προωθήσουμε τη συνεργασία, το διάλογο, χωρίς να δημιουργήσουμε τα σχέσεις προσπαθώντας να βρούμε λύσεις. Προσπαθούμε να ενεργούμε ε, πάντα έχοντας κατά νου το κράτος δικαίου δημιουργήθηκαν κάποιες ε, αστυνομικές αρχές οι οποίες σιγά σιγά οριμάζουν, πράγμα το είναι θετικό όσον αφορά τη λειτουργία τους. Εάν θέλουμε να υπάρξει σταθερότητα, θα πρέπει και σε επίπεδο αστυνομίας να γίνει σωστή ε, στελέχωση για να λειτουργούν σωστά. Θα πρέπει να ξέρουν πώς να λειτουργούν για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις κρίσεις. και θα πρέπει να υπάρχει και μεταξύ του συνεργασία. Όπως σας είπα, και σε διεθνές επίπεδο συνεργαζόμαστε για να δούμε αν μπορούν αυτές οι αστυνομικές αρχές να λειτουργήσουν σωστά και από μόνο τους. Και πρέπει να σας πω ότι η αστυνομία δεν δουλεύει μόνη της για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να δημιουργεί σχέσεις και δίκτυα με τους άλλους. Αυτό το λέγω από την μεγάλη εμπειρία που έχω στην τομέα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσει να εκδιωχθεί το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά. Αυτό είναι θετικό, αλλά βεβαίως όλο περισσότερο οργανωμένος είναι ο μεν, τόσο περισσότερο αντιδρά Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία και συνδρομή. Όχι διότι εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Κοινότητας πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό, αλλά γιατί το λένε οι εταίροι μας σε τοπικό επίπεδο, διότι όπως λέγουν εποφελούνται από συνεργασία που τους βοηθά για να θεσπίσουν κάτι το δύσκολο σε αυτό το πολιτικό ευαίσθητο περιβάλλον. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι για αυτές για να μπορέσουν να επιληθούν οι πολιτικές προκλήσεις και να προχωρήσει η κατάσταση θετικά, πρέπει να προχωρούμε χωρίς να προσπαθούμε να βρίσκουμε πάντα εξηγήσει που να αρμόζουν στις απόψεις των Γάλλων των Ιταλών, αλλά λύσεις οι οποίες να αρμόζουν στην τοπική κατάσταση που επικρατεί στη Βοσνία Σγοβίνη. Και αυτό είναι ένα στιγμίο ισχυρό, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμούν όχι μόνο σε επίπεδο δημιουργίας αυτών των διοκτικών αρχών, αλλά και σε όλες τις συζητήσεις που είχα και στο παρελθόν και στην Πανιαλούκα και στην Σερβική Δημοκρατία και σε πολλούς άλλους. Και βεβαίως, όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολιτικά και κομματικά κριτήρια όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκαν κάποιες τελευταίες διώξεις που έγιναν τα οποία εμείς δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Όχι διότι ε, πρέπει να... διότι εμείς έχουμε στόχο να φέρουμε σε πέρας μια τεχνική αποστολή. Όχι ότι θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά πρέπει να είμαστε αμέτωχοι. Και όπως και σε όλες τις περιπτώσεις τις οποίες ενεργούμε επιτόπου, όπως έγινε στο παρελθόν στα πλαίσια αποστολών που είχαν στα πλαίσια του ΟΗΕ, σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους τεχνική αποστολή θα πρέπει να έχετε πάντα μία πολιτική ε, κάλυψη και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο με την κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο έχουμε επιτύχει. Είμαστε πάρα πολύ ε, κοντά με τους εταίρους, τους τοπικούς πολιτικούς επιτόπου και βεβαίως με όλους τους συνομιλητές μικρούς ή μεγάλους, της είπα ή κάποιους άλλους, με τους οποίους πρέπει να ενεργούμε. Εάν δεν είχαμε ένα τέτοιο πνεύμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα υπάρχουν προβλήματα που ξεπερνούν κάποιες χρονικές περιόδους και πρέπει να επιμείνουμε. Όντως, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα ε, μειονεκτήματα και τα ε, πλεονεκτήματα που πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να δούμε τι κάνουμε με τα οικονομικά εγκλήματα, για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, για θέματα οικονομικά, αλλά πρέπει να έχουμε και τους κατάλληλους πόρους. Ο συνάδελφος Σίπα Σικολούιτς αναγνωρίζει ότι όλες, τις, όλες τις συζητήσεις που έχει με μένα και με άλλους λέγει ότι ο οργανισμός του, το οποίο δημιουργεί το 2003, ακόμη πρέπει να σημειώσει πρόοδο. Και το σύστημα ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει παγιωθεί δεν έχει αναπτύξει την ταχύτητα που του χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν ελλείψεις, μειονεκτήματα, τα οποία σιγά σιγά ε, πρέπει να ξεπεράσουμε και όχι μόνο με την ε, βοήθεια της ε, αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα νοικονομική συνδρομή αλλά και με διάφορα προβλήματα, τα οποία, προγράμματα τα οποία αφορούν την προστασία των ματήρων, την ε, διασυνοριακή συνεργασία και διαχείριση διασυνοριακών προβλημάτων για το ΟΝΑ σάνα. Θα πω ότι το ούνα σάνα είναι ένα παράδειγμα και μπορώ να σας δώσω ένα κατάλογο νέων τέτοιου είδους παραδειγμάτων που δεν θα σας δώσει νέε προφορίες. Απλώς πρέπει να σας πω ότι δεν ασχολούμαι μόνο με το Ουνασάνα. Πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση την οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε για να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο διότι πάντα προσπαθούμε να βρούμε αυτή την λύση. Τώρα, πώς μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες και πώς να αξιολογείται. Υπάρχει βελτίωση. Στην περίπτωση της ε, Βοσνίας Εσεργοβίνης, βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν δραστηριότητες θα θέλαμε να είναι πιο συντονισμένες ακόμη και σε επίπεδο επίσημο. Υπάρχουν όμως εξελίξεις ε, που θα πρέπει να υπάρξουν. Θέλουμε να έχουμε περαιτέρω συντονισμό των προσπαθειών που καταβάλουμε. Και αν δεν κάνω λάθος και δεν μου πει τίποτα συμπληρωματικό πρόεδρος τώρα, νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις. Euh, Ευχαριστώ. θα υπάρξει μια αποστολή της υποεπιτροπής μας που θα πάει στο Σαράγεβο για την, και για την Αλτέα αλλά και για την αστυνομική αποστολή. Πέρα από τα πολιτικά προβλήματα που αναφέρθηκαν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπατε εσείς ε, για την αποστολή σας. Ο κ. Ντεμαγνιάκα θα συζητήσει, συζητάει νομίζω με τον ε, εισηγητή μας για το κοσφοπέδιο. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Θα παραμείνουμε ε, σε επαφή γιατί η στρατιωτική και η πολιτική αποστολή στα Βαλκάνια είναι πολύ σημαντική ε, δράση της ΚΠΑ. ΚΠΑ. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα της Λιβύης. Σας ζητάω δύο λεφτά διάλειμμα. Merci de reprendre place. Παρακαλώ καθίστε. Να σας πω δύο λόγια. Είχαμε βάλει στην ημερήσια διάταξη μία συζήτηση για την έκθεση του συναδέλφου Γκουαλτιέρη για την ΕΚΠΑ μετά τη συνθήκη της, Λισαβόνας. Σε συμφωνία με τον Ρομπέρτο αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση γιατί η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών παρατάθηκε είχατε μέχρι αύριο για τροπολογίες και θα έχουμε μία ειδική συζήτηση στο Στρασβούργο στην επόμενη Ολομέλεια για την έκθεση αυτή. Μία συζήτηση πολύ πιο λεπτομερή. Ε, σήμερα δεν υπάρχουν και νέα στοιχεία σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα και όλες οι τροπολογίες δεν έχουν ακόμα κατατεθεί. Ε, και ο Ρομπέρτο βέβαια δεν έχει δει το σύνολο των τροπολογιών. Τον ευχαριστώ λοιπόν που δέχτηκε την αναβολή. Θα κάνουμε αυτή την εκτεταμένη συζήτηση στο Στρασβούργο στην επόμενη Ολομέλεια στις 4 Απριλίου. Περνάμε τώρα ε, στο, σε ένα σημείο επικαιρότητα. Είναι πιο σημαντικό να το δούμε αυτό. Ε, ήταν το κοσφοπέδιο θέμα επικαιρότητα, αλλά και η Λιβύη, γιατί οι εξελίξει στη Λιβύη είναι καταιγιστικέ και δυστυχώ δεν είναι, δεν είναι δεν θεωρούμε πια ότι είναι δεδομένη η εξέλιξη βραχυπρόθεσμα όπως θέλουμε. Την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ε, εξέδωσε ένα ψήφισμα για τη Λιβύη που έχει κάποιες συστάσεις, προτάσεις ε, και για πολιτικό, σε πολιτικό επίπεδο την αναγνώριση του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου, την δημιουργία μιας περιοχής απαγόρευσης πτήσεων, καθώς και τη δυνατότητα για την ε, ύπατη εκπρόσωπο να μελετήσει και να διερευνήσει τη χρήση των ε, μέτρων ε, ΚΠΑ με βάση το ψήφισμα 1970 του ΟΗΕ για το εμπάργκο στη Λιβύη ε, στις 11 συνεδριάζει εκτάκτος, συνεδριάζει εκτάκτος μάλλον το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο λέει για να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό τα κράτη-μέλη θα μελετήσουν όλες τις απαραίτητες ε, εναλλακτικές λύσεις εφόσον υπάρχει μια σαφής νομική βάση και δεδομένης της ε, ε, ανθρωπιστικής ε, ανάγκης ε, θα υπάρξει υποστήριξη της ανθρωπιστικής προσπάθειας. Ε, είναι ένα αόριστο κείμενο, ε, πολλά στοιχεία ανοιχτά. Σήμερα οι δυνάμεις του Καντάφη έχουν ανακτήσει το χαμένο έδαφος και οι εξεγερμένοι στρατιωτικά βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Οι συζητήσεις για τη δημιουργία μιας περιοχής απαγόρευσης πτήσης ε, συνεχίζονται. Οι συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Καλό είναι να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ τον κύριο Ποπόφσκι που, μας, που ήρθε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει αποτίμηση του Συμβουλίου της Παρασκευής, των διαμηθών του Συμβουλίου την Παρασκευή δηλαδή. Θέλουμε και εμείς και ο συνάδελφο και ο, κατηγορ, και ο, συγγνώμη, ο μιλητής μας να επικεντρωθούμε στα θέματα της ΚΠΑ. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτικά θέματα. Έτσι μπορείτε να τα θέσετε εσείς, αλλά μπορείτε να μην λάβετε απάντηση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, θα δοθούν αύριο από τον πρόεδρο Φαν ε, σε μια ε, συνέντευξη τύπου ανοιχτή για όλους τους βουλευτές. Θέλω να μιλήσουμε, να επικεντρωθούμε λοιπόν στα θέματα ασφάλειας και στα θέματα άμυνας. Κύριε Ποπόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πριν περάσω στα θέματα ασφάλειας ε, στη Λιβύη, θα ήθελα να υπενθυμίσω τη γενική μας προσέγγιση. Υπάρχει τώρα μια κοινοτική προσέγγιση γενικά για την Βόρεια Αφρική. Ε, τα μέτρα της ΚΠΑ, ε, τα μέτρα της ασφάλειας είναι τμήμα του ευρύτερου πακέτου. Όπως βλέπετε και στην ανακοίνωση που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί γίνεται λόγος για διάφορα θέματα, όπως η πρόσβαση στην αγορά και η μετακίνηση του εργατικού δυναμικού, ε, πρόσβαση που θέλουμε να προσφέρουμε στους νότιους γειτονές μας. Φυσικά αυτή τη στιγμή ανησυχούμε για τα πρόσφατα γεγονότα, για την εξέλιξη, τις εξελίξεις στη Λιβύη. Θα ήθελα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια καταρχήν. Οι βασικές μας προτεραιότητες μέχρι στιγμής ήταν η εκένωση των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων από την ε, Λιβύη ε, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στα σύνορα της Λιβύης έχουμε εκενώσει χιλιάδες ανθρώπους. Ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν λειτουργήσε ομαλά και έδωσε προστιθέμενη αξία ανταλλάξαμε πληροφορίες πολύ γρήγορα και χρησιμοποίησαμε τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους σπόρους που είχαμε. Ε, υποστηρίζαμε την, τις προσπάθειες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ ως υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ε, κινητοποιώντας το στρατιωτικό προσωπικό και ε, χάρη σε ένα πυρήνα ε, συντονισμού όπως το λέμε. Επίσης έχουμε έναν αξιωματικό ε, συνδέσμου στην αποστολή συντονισμού στην την Ισία, επίσης ένα άλλο αξιωματικό ε, στη Μάλτα για συντονιστικό έργο. Από τα όσα μαθαίνουμε από την Γενική Διεύθυνση και τον ΟΗΕ είναι ότι υπάρχει προσωπικό για να εκενώσουν τα άτομα τα οποία φτάνουν από τη Λιβύη στην Ισία. Θα συνεχίσουμε το συντονισμό πιο ενισχυμένα όμως. Όλα αυτά δεν είναι γνωστά. Γι' αυτό επικοινωνούμε, για να εξηγήσουμε στον τύπο και στα ΜΜΕ τι κάνουμε από την αρχή της κρίσης. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι, το πιο, η πιο άμεση ας πούμε, απόκριση είναι η εκένωση. Επίση, επίσης η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ήταν τα δύο πρώτα πράγματα. Κάνουμε κάποιο σχεδιασμό για να δούμε τι εναλλακτικέ λύσει έχουμε στα πλαίσια της ΕΚΠΑ ε, στη Βόρεια Αφρική. Το ΝΑΤΟ κάνει την ίδια προσπάθεια όπως ξέρετε και ξεκινήσαμε κι εμεί, Πολύ πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας. Οποιαδήποτε δράση ΚΠΑ θα εντάσσεται στο συνολικό πακέτο μέτρων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι εξετάζοντας τις εναλλακτικέ λύσεις για την προστασία των ε, άμαχων πληθυσμών ακολουθεί τρεις ε, αρχές ε, την ανάγκη, την νομική βάση και την υποστήριξη της περιοχής. Είναι ίδια η προσέγγιση με του ΝΑΤΟ. Οι Υπουργοί Άμυνα συναντήθηκαν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και συμφώνησαν με τις ίδιες αρχές. Αρχές που θα καθοδηγήσουν τις δικές τους δραστηριότητες, οι οποίες είναι να εξελίξει ξεκινήσαμε έναν προσεκτικό σχεδιασμό πιθανών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βραχυπρόθεσμα, δράσεις δηλαδή ΚΠΑ ε, για την κρίση στη Λιβύη, καθώς και μεσοπρόθεσμες μακροπρόθεσμε μακροπρόθεσμες ε, δράσεις για την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών και στις τρεις χώρες, σε Λιβύη, την Ισή και Αίγυπτο, καθώς και δράση στον τομέα της ασφάλειας. Βραχυπρόθεσμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που ανέφερα, θα είναι να υποστηρίξουμε περισσότερο για, με σκοπό την εκένωση και υποστήριξη της ανθρωπιστικής προσπάθειας, ε, μια στενή ας πούμε θαλάσσια γέφυρα, ε, βοήθεια σε μηχανικό επίπεδο, ιατρικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο, επίσης μέτρα για την υποστήριξη της εφαρμογής του εμπάρκου όπλων που επιβλήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παρότι και από νομικής απόψεως είναι σαφές ότι η εφαρμογή του εμπάρκου οποιοδήποτε οργανισμό ε, θα απαιτήσει άλλη εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σχεδιασμός είναι λοιπόν ψηλαφιτός, προσεκτικός. Δεν προδικάζουμε λοιπόν τις, απόφυσ, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ε, κάνουμε σύγκριση των ε, προσπαθειών μας με το ΝΑΤΟ με διαφανή τρόπο δηλαδή. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν ε, την ευαισθησία των σχέσεων με το ΝΑΤΟ, ενημερώνονται, ε, λειτουργούμε με διαφάνεια. Δεν θέλουμε να υπάρξουν επικαλύψεις, θέλουμε να εστιάσουμε στη δουλειά που μπορούμε εμείς να κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και να επιφέρει προστιθέμενη αξία για να αυξήσει και το δυναμικό μας αλλά και την εμπειρία μας. Και να χρησιμοποιήσουμε και το δυναμικό μας αλλά και την εμπειρία μας. Ε, η συζήτηση τώρα για την ζώνη απαγόρευσης πτήσεων γίνεται και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι θα καταλήξει και θα υλοποιηθεί σύντομα. Γιατί όλοι περιμένουν μια καθαρή εντολή. Η υποστήριξη, αλλά και την υποστήριξη της περιοχής. Οι, οι Άραβες ηγέτες ζήτησαν την δημιουργία μιας τέτοια ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Αλλά αυτό δεν προδικάζει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είναι ακόμα διστακτικά. Ε, οι Υπουργοί Εξωτερικών του G8 συναντήθηκαν χθε στο Παρίσι και είμαι σίγουρος ότι αυτό ήταν από τα βασικά θέματα της συζήτησής τους, όπου η εκπρόσωπος συμμετείχε και αυτή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απαιτείται κάποια δράση. Εμείς εκεί μπορούμε να επιφέρουμε τη θεμενή αξία. Κατά τη γνώμη μας. Και για τις τρεις χώρες, όταν υπάρξουν συνθήκες εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την ε, πραγματογνωμοσύνη μας για τη διαχείριση της μεταβατικής ε, κατάστασης. Δηλαδή, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ε, ασφάλειας, της δικαιοσύνης, κράτος δικαίου. Αυτό το κάνουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην Παλαιστίνη, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ινδονησία ακόμα. Μπορούμε να το προσφέρουμε λοιπόν και στη Βόρεια Αφρική, θα πρέπει όμως να το ζητήσει η περιοχή σαφώς. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Όταν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό και το συζήτησα και με το τμήμα σχεδιασμού και με το στρατιωτικό προσωπικό, εμείς είμαστε διαφορετικοί από τον ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να συγκριθούμε ακριβώς με τον ΝΑΤΟ. Ε, στο επιτελείο του ΝΑΤΟ έχετε χιλιάδες σχεδιαστέ που ασχολούνται με τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Εμείς έχουμε καμιά δεκαριά άτομα τα οποία ασχολούνται με το σχεδιασμό. Επομένως είμαστε σε άλλη κλίμακα του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά την μια αποστολή στα πλαίσια της ΚΠΑ για την παρακολούθηση και συμβουλή για θέματα μη στρατιωτικά και για θέματα διοίκηση, ας πούμε, μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Μπορούμε να βασιστούμε στην εμπειρία που έχουν κάποια κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο των ε, ενόπλων δυνάμεων, την ε, μεταβατική δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, πάρα πολύ σημαντική πρόκληση που έχουμε δει και σε άλλες χώρες τα τελευταία 20-25 χρόνια και βεβαίως ε, το τομέα της ασφάλεια και μεταρρυθμίσεις για την ασφάλεια. Αλλά αυτά είναι μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η εκένωση και τα ανθρωπιστικά θέματα. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, να σταματήσω εδώ ε, και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις και να ακούσω σχόλια. Ευχαριστώ. Πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο Αν μου επιτρέπετε, θέλω να εκφράσω κάποιες απογοητεύσεις, κάποιες δυσαρέσκειες που έχουμε συσσωρεύσει. Γιατί ακούω, εντάξει, τις επιτυχίες που είναι αναφυσβήτητες. Θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν οι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αφορά την εκένωση και την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό κανένα δεν το αμφισβητεί. Έγινε δουλειά με καλό τρόπο και όπω υπενθυμίσατε κι εσεί ε, δεν έχει τελειώσει και όλοι είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Κατά τα λοιπά τώρα, μιλάμε για συνετό, λέει, σχεδιασμό. Μας μιλάτε για μέσο μακροπρόθεσμη προσπάθεια να συνοδεύσουμε την προσπάθεια α, μετάβασης. Αλλά στη Λιβύη δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε στο τι γίνεται τώρα. Ε, χαίρομαι που ξεκίνησαν σχεδιασμός τουλάχιστον, έστω και συνετός, γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Αλλά ε, σε όλα αυτά τα κατεπήγοντα θέματα της Λιβύης, πώς μπορεί να απαντήσει όταν εμείς στραφούμε προς τους συμπολίτε μας, πάντα μας ρωτάνε τι κάνει η Ευρώπη. Άλλοι φορείς, ιδίω οι ΙΠΑ, έδειξαν μεγάλο σκεπτικισμό απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή προσπάθειας που να έχει την πτυχή ασφάλεια και άμυνα. Ε, όταν εγώ τους λέω συνετός σχεδιασμός, νομίζω θα μας καταλάβουν οι συμπολίτε μας. Ξέρω βεβαίω ότι το ΝΑΤΟ έχει πολύ, πολύ πιο σημαντικά μέσα, αλλά και εμεί έχουμε τα δικά μα. Υπάρχει μία θαλάσσια αποστολή κατά της πειρατείας ε, που εκτείνεται χιλιάδες χιλιόμετρα τις ακτές μας. Γιατί δεν μπορεί η, να κάνει μια θαλάσσια αποστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις δικές της ακτές. Δεν καταλαβαίνω όταν έχουμε πολύ πιο μακρινές αποστολές. Καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να μα τα αποκαλύψετε όλα, αλλά θέλω περισσότερε ενδείξει. Όλα τα στοιχεία και τα εργαλεία τα οποία έχουμε, τα οποία έχει η κυρία Άστον στη διάθεσή τη. Χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού, για να δούμε όλε τι δυνατότητε που έχουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, και κάποιε προποθέσει, όπω είπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά έχουμε διάφορε εναλλακτικέ λύσει ε, στη διάθεσή μα. αυτή η ορολογία σκεπτική και προσεκτική σχεδίαση, σχεδιασμός. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμπεριλαμβάνει. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν ε, για αυτή την ε, δυσαρέσκεια που αισθανόμαστε και αυτό το σκεπτικισμό. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, έγινε μια πλούσια συζήτηση, Ψηφίστηκε ένα ψήφισμα. Θα ήθελα να τα πείτε όλα αυτά στην ύπατη εκπρόσωπο. Ε, οι απαντήσει που μα δώσατε δεν είναι στο ύψο των προσδοκιών μα, αλλά οι δικέ μα προσδοκίε είναι σε ευθεία γραμμή με τι προσδοκίε των συμπολιτών μα. Αυτά. Ο κύριο Γκάλερο, επόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Παπόφσκι. Και εγώ συμμερίζομαι την δυσαρέσκεια του Προέδρου της Επιτροπής μας Διάβασα όλα τα έγγραφα τα οποία ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις τελευταίες ημέρες, τα σχόλια του Πρόεδρου Φαρόμπαϊ, τη δήλωση της Βαρόνης Άστον, το κείμενο της Αραβικής Λίγκας και τα συμπεράσματα τα οποία εξαγάγω είναι ότι η Λέδη πολύ απλά δεν θέλει να μας παρουσιάσει τις δυνατότητες που έχουμε. Θέλει τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή τον οποίο έχουμε και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα. Διαφορετικά θα έπρεπε να κατανοήσει το ρόλο της. Κοιτώντας τις αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι έχουμε ανοιχτές όλες τις δυνατότητες Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι ομάδες εργασίας που συμμετέχουν σε αυτόν τον ε, σχεδιασμό, το prudent planning στην παρούσα φάση. Θα με ενδιαφέρει αυτό αφενός. Αλλά αν έχουμε ανοιχτέ όλες τις δυνατότητες και θέτουμε τρεις όρους, αυτό που ερωτώ είναι το εξής. Θεωρείτε ότι υπάρχει αποδεδειγμένα ανάγκη παρέμβαση στην δεδομένη και της κατάστασης της ανθρωπιστικής. Στη Λιβύη θεωρείται ότι, η υποστήριξη, ότι υποστήριξη από την περιοχή, από την περιφέρεια και πώς έχουν έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για μια ζώνη απαγόρευσης ενέργειας ε, κυκλοφορίας, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν συμφωνούν τα κράτη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι είναι σαφής η θέση της Αραβικής ε, Λίγας. Δεν θέλει foreign intervention, ε, ξένη παρέμβαση. Αυτό αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο, αλλά στην επόμενη παράγραφο ε, απαιτεί άμεσα αυτά no-fly zone. και δεν ερμηνεύει μια τέτοια παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ως foreign intervention. Αυτό θεωρώ ότι υπάρχει υποστήριξη από την περιφέρεια όταν αναφέρεται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφαρμόσουν άμεσα μια απαγόρευση ενέργειας κυκλοφορίας. Μα τι θέλουμε ε, πλέον από την περιοχή. Πώς θέλουμε να αντιδράσει, πόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να αντιδράσει η περιφέρεια. Θέλει να κρυφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την Αφρικανική Ένωση. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς λοιπόν πώς τοποθετούνται τα κράτη-μέλη στο... για το no-fly zone. Με ονόματα αν γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Γκουατιέρη. Ευχαριστώ. Ένα τεχνικό σχόλιο θα ήθελα να πω. Όσοι κάνουν το library briefing να γράφουν αυτό που έγραψε το ψήφισμα που ψήφισε το Κοινοβούλιο, που είναι διαφορετικό από αυτό που γράφεται εδώ για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου λέει ξεκάθαρα ότι η non-flying zone είναι μια δυνατότητα που θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί μόνο αν υπάρξει εντολή του ΟΗΕ. Αυτή λοιπόν η ζώνη απαγόρευση πτήσεων ε, εγκαθιδρύεται μόνο υπό αυτόν τον όρο. Αυτό ψηφίστηκε την Ολομέλεια. Πολύ ωραία. Μετά από αυτά, θέλω να σας πω ότι το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Και η σύνεση που εκδηλώνεται από το Συμβούλιο και από την ύπατη εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό βέβαια Συμβούλιο και από την ύπατη εκπρόσωπο, είναι βάσιμη. Έχει νόημα. Συμφωνώ με τις τρεις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. για να ξεπεράσουμε το ψήφισμα του 1970. Δηλαδή, περιφερειακή υποστήριξη, που σημαίνει και υποστήριξη από την Αφρικανική Ένωση, ξεκάθαρη νομική βάση, και συγκεκριμένα στοιχεία για το τι συμβαίνει επί τόπου. Λείπουνε όμως αυτά τα στοιχεία, πρέπει να το πούμε. Και από αυτόν χρήσιμο θα ήταν να μας πει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση, το Situation Center, να μας δώσει κάποια στοιχεία, κάποια γεγονότα. Γιατί αυτό που με ανησυχεί σε αυτή την κρίση για τη Λιβύη είναι ότι πέρα από κάποια νούμερα, τα οποία είναι λίγο απίθανα που μας δίνουν διάφορες ε, εφημερίδες ε, οι οποίες αναφέρουν πηγές από τις χώρες του κόλπου. Τελικά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει επί τόπου. Η, Αραβική, ε, η, η Σαουδική Αραβία λέει ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί δεν οδήγησαν σε θύματα σε πολλές πόλεις. Δεν, δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν δύο στρατοί, δηλαδή οι οποίοι αντιπαρατίθενται ή έχουμε μια, ένα πόλεμο ας πούμε πραγματικό με δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες θύματα. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα θύματα. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις δεσμευτικές για αυτό το non-flight zone που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι εκ των όνου κάνευ, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, η κατάσταση επιτόπου να είναι τέτοια που να το καθιστά αναγκαίο, ούτω ώστε να υπάρξει μαζική παρέμβαση. Αυτό σημαίνει βομβαρδισμό λοιπά. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δημιουργούμε ένα στρατιωτικό ε, εξοπλισμό και μηχανισμό τρομερά ε, επαχθή. Ότι μπαίνουμε στην περιοχή ουσιαστικά. Αυτή η απουσία λοιπόν ειδήσεων για το τι συμβαίνει στη Λιβύη μας αποπροσανατολίζει και δεν μπορούμε να πάρουμε πολιτική θέση. Ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, και δικαιολογούν και κάποιες βιαστικές, ας πούμε, απόψεις του Κοινοβουλίου. Για να μπορούμε να έχουμε σοβαρές απόψεις για την εξωτερική πολιτική και να μην είμαστε μόνο αντιχείο της α, κοινή γνώμης, θα πρέπει, για να το κάνουμε αυτό, να έχουμε και τα στοιχεία στα χέρια μας. Ε, όμως, σύνεση δεν σημαίνει αδράνεια, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω ότι θέλει να πει και ο πρόεδρος Ντόνζο. Γιατί σύνεση για το θέμα του πολέμου δεν σημαίνει ότι περιοριζόμαστε μόνο στην εκένωση και στον επαναπατρισμό. Και με το σημερινό ψήφισμα του ΟΗΕ έχουμε μεγάλο περιθώριο για μεγάλες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να αφορούν τον τρόπο ενεργοποίησης του εμπάργου Βέβαια, υπάρχει και ένα πρόβλημα νομικής βάσης. Μπορεί επίσης να προβλέψει και στοιχεία της ΚΠΑ, όπως ακριβώς ε, λέει και το... και μηχανισμού και εργαλεία της ΚΠΑ, όπως λέει και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Επίσης, η Λιβύη είναι πολύ περίπλοκη α, χώρα. Έχει τρεις βασικές φυλές ε, που κάνανε μια συμφωνία γύρω από τον Καντάφη. Αυτή η ενότητα των φυλών έχει τεθεί σε αμφισβήτηση αν υποστηρίξουμε αυτούς τις βενγκάζεις, μπορεί παραδόξως να ενισχύσει την ενότητα των φυλών. Αλλά όμως θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα πολιτικός χώρος ε, κατάπαυσης του, πυρός, ας πούμε, ούτως ώστε να ξεκινήσει αυτή η ενδιάμεση φάση, ας πούμε, η, φάση της μετάβασης. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει αυτή τη δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να κατακαιρματιστεί τώρα σε μια συζήτηση για, στρατιωτικέ για στρατιωτικές λύσεις που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Όχι. Θα αποφασίσουμε. Θα περάσουμε στο εμπάργο. Θα παγώσουμε τα οικονομικά στοιχεία ε, των μελών του καθεστώτος. Κάτι που ζητάει η Αφρικανική Ένωση. Θα ξεκινήσουμε μια πολιτική πρωτοβουλία που θα βασίζεται όμως σε πραγματική γνώση των πραγματικών δυνάμεων που δρούν στη Λιβύη Πρέπει να έχουμε αυτές τις γνώσεις για να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, κυρία Μπράτνερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για το γεγονός ότι ήρθατε. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά να κάνετε στην παρούσα φάση. Υπάρχει και η Ιαπωνία στην ημερήσια διάταξη και στην παρούσα φάση δεν ξέρουμε πού να ξεκινήσουμε ουσιαστικά. Γι' αυτό που, για το ερώτημα του ποια είναι τα γεγονότα, ποια είναι τα περιστατικά Ελπίζουμε να έχουμε πιο να έχετε πιο πολλές πληροφορίες από ό,τι εμείς, γιατί στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι ο κίνδυνος είναι η μπεγάζη να περικυκλωθεί και αν ε, διαρκέσει η κατάσταση μερικές ημέρες να γίνει αιματοχυσία, να καταλάβει την πόλη ο Καντάφη. Και το θέμα που ανακύπτει είναι τι πρέπει να κάνουμε τώρα, όχι σε επίπεδο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Μιλάμε σε επίπεδο ημερών. Ιδάλλως δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση κατά του Καντάφη και πώς θα τον υποστηρίξουμε. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη. Στην περίπτωση αυτή ε, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο κύμα αντιφρανούντων. Αλλά στην περίπτωση αυτή τι θα έχουμε δηλαδή μια πολιτική ε, η οποία θα ανταποκρίνεται στις αρχές μας για την ε, ανθρώπινα δικαιώματα, γίνομαι κάπως κοινική. Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά μας και ε, επίσης κατά πόσο θα συνεργαστείτε με την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι και αυτός ένα πολύ σημαντικός παράγοντας. Η τοποθέτηση της Τουρκίας για την απαγόρευση ενέργειας κυκλοφορίας και το θέμα επίσης μη, πέρα από την ε, Λιβύη αναφέρατε την δυνατότητα αποστολής, αποστολών κρατούς δικαίου στην Τινησία και στην ε, Αίγυπτο. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου γιατί για παράδειγμα ε, υπάρχει και αυτή η αποστολή κρατούς δικαίου στο Ιράκ η οποία δεν στέφθηκε ακριβώς με επιτυχία. Πώς λοιπόν θα οργανωνόταν μια τέτοια αποστολή και πώς θα διασφαλίζαμε ότι θα εντάσσονταν σε ένα συνολικό πλαίσιο θα, ότι θα είχε αρμοδιότητα και ο επικεφαλής της αποστολής. Νομίζω ότι θα έπρεπε εξ αρχής να δράσουμε πολύ συντονισμένα για να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες όπου θα έχουν δοθεί τα κονδύλια και θα υπάρχει αποστολή αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιος επικεφαλής ο οποίος θα είναι υπεύθυνο και επίση μια εκτίμηση αν θέλετε για τον Παχρέιν. Κυρία Λούζινγκ, ναι σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκαουτιέρη, τον Γκουαλτιέρη για τις ε, παρατηρήσεις του. Με πολλές από αυτές συμφωνώ. Είχαμε σήμερα το πρωί τη συζήτηση στο Κωσυφοπαίδιο. Βλέπουμε πώς έχει η κατάσταση στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Έμα ε, κάποια μαθήματα θα πρέπει να εξαγάγουμε. Καταλαβαίνω την ανάγκη να βοηθήσουμε. Καταλαβαίνω την αιματοχυσία, την δικτατορία του Καντάφη. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά δεν μπορούμε να ακολουθούμε το δόγμα ότι πρώτα θα υπερβολήσουμε και μετά θα κοιτάξουμε τι έγινε. Γιατί πολύ απλά δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πρέπει να αναλύσουμε ποιες δυνάμεις, υπό ποιους όρους και με ποια μέσα μπορούμε να υποστηρίξουμε και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μία, ένα σχεδιασμό μακροπρόθεσμο για το πώς έχει η κατάσταση μετά την παρέμβαση γιατί αυτή η κατάσταση θα επικρατήσει επί δεκαετίες, πολλές δεκαετίες θα μείνει έτσι η κατάσταση μετά Ε, να περάσω σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα και για την απαγόρευση ενέργειας κυκλοφορίας. Ε, πολλές φορές το ακούσαμε και πολλές και διαφορετικές είναι οι απόψεις που επικρατούν πολύ και ο Υπουργός Άμυνας Γκέιτς πιστεύουν ότι σε περίπτωση απαγόρευσης και σε περίπτωση που εφαρμοστεί η απαγόρευση θα υπάρξει πόλεμος. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε ε, του Strategic Fit Forecast προειδοποιούν και διαμηνύουν ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του Καντάφη βρίσκονται σε πόλεις με μεγάλους πληθυσμούς και έτσι ε, σε περίπτωση που υπήρχε τέτοια παρέμβαση θα υπήρχαν πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων. Τα στρατεύματα του Καντάφη ουσιαστικά δεν θα αποδυναμόντουσαν σε περίπτωση απαγόρευσης ενέργειας κυκλοφορίας. Συμφωνείτε με την εκτίμηση αυτή. Αν όχι, γιατί. Το Ίδρυμα για τις Έρευνες Ασφάλειας ε, ε, δημοσίευσε μία ανάλυση η οποία ε, υποστηρίζει ότι μία στρατιωτική παρέμβαση βάσει της ευθύνης προστασίας μπορεί να γίνει χωρίς και χωρίς εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Ερωτώ, συμφωνείτε? Μία ερώτηση για την ανθρωπιστική βοήθεια συχνά παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι μια βασική, ένα βασικό καθήκον της ε, αποστολίας ε, της Frontex Ερμής 2011 να υποστηρίξουν ε, την πρόθεση των προσφύγων στις χώρες προέλευσης. Συμφωνείτε και πώς αυτό επιδρά και αφορά τους πρόσφυγες της Λιβύης. Οι πρόσφυγες θα επιστραφούν στον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο δεν θα έπρεπε να δεχτούμε όλους τους πρόσφυγες από τη Λιβύη και να αναπτύξουμε ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστώ. Και οι πολιτικές ομάδες έλαβαν το λόγο Κατά τη διάρκεια του πρώτου αυτού γύρου ερωτήσεων θα δώσω το λόγο στον κύριο Ποπόφσκι και μετά θα επανέλθω. Θα ήθελα πριν να σα δώσω το λόγο να κάνω τρεις παρατηρήσεις όσον αφορά αυτή την έννοια της με μετριοπάθεια. Είπε κανεί ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, από πολιτική πλευράς και κυρίως πριν να αναλάβουμε όποια δέσμευση. Επίση, ε, ελέγχθη κάτι για τον ε, προσεκτικό σχεδιασμό. Τι σημαίνει αυτό. Κάπως περιοριστικό. Ή προετοιμαζόμαστε και σχεδιάζουμε σωστά ή όχι. Επίσης, η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Πριν ε, να συσταθεί μια τέτοια ζώνη θα πρέπει να γίνουν μεγάλες νέες χερσαίες ε, καταστροφές. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε για την Βοσνία D-Night Flight, η οποία έγινε χωρίς να υπάρχει απαραίτητο να γίνει καμία χερσαία επιχείρηση. Το 95 ε, επίσης θα υπενθυμίσω μία άλλη επιχείρηση. Στη Βοσνία όμως 93-95 πρέπει να πω ότι με επιτυχία εφαρμόστηκε αυτή η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Επίση, συμφωνώ αυτό που η κυρία Ζήν και αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση. Η ζώνη υπαγορευτήσεων σίγουρα δεν θα επιλύσει όλα ή ένα μέρος των σοβαρών στρατιωτικών προβλημάτων που τίθεται επί τόπου και οδηγούν σε διάφορες επιχειρήσεις από, την, ε, από τον ε, στρατό ξηράζοντα τα βαρέα πυρομαχικά. Πιστεύω λοιπόν ότι από ιστορικής πλευράς, επειδή ακούστηκαν και διάφορα επιχειρήματα τα οποία είναι ασαφή, πρέπει να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ίσως θα πρέπει να κάνω μία ε, διευκρίνηση για αυτό το prudent planning. Είναι τρόπος να αρχίσει κανείς μία διαδικασία χωρίς να την επισημοποιήσει. Και αυτό που είναι Σημαντικό είναι να πούμε ότι εσείς ε, είστε ίσως ε, ειδικοί σε θέματα στρατιωτικού σχεδιασμού, υπάρχουν κάποιες έννοιες τις οποίες χρειάζεται. Εμείς δεν θελήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο επισήμως, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό με προσοχή. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη Καταλαβαίνω τον σκεπτικισμό και την απογοήτευση κάποιων, έτσι όπως εκφράστηκε από κάποιος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία. Ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλυφθεί κάποια πολύ ισχυρή δράση εκεί. Ξέρω ότι συνεδρίασαν πες το βράδυ στο Παρίσι, πρέπει να πω ότι κάποιοι παραμένουν σιωπηλοί σε επίπεδο ε, Συμβουλίου Ασφαλείας. Δύο μέλη είναι αντίθετα ώστε να υπάρξει μια, ένα ψήφισμα ισχυρό. Ξέρω ότι υπάρχει μια πρόταση νέου ψηφίσματος εκ μέρους της Γαλλίας για να ξεπεραστούν τα πλαίσια της ε, απόφασης 19-17, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή δεν υπάρχει ομοφωνία δεν μπορεί να δοθεί τέτοιου είδου εντολή και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει με αφιστικό τρόπο χωρί να υπάρχει νέα εντολή. Αυτό είναι σαφές. Θα ήθελα τώρα να τονίσω το εξή. Βεβαίω υπάρχει διαφορά μεταξύ της ε, σχεδιασμού που γίνεται σε επίπεδο ΟΗΕ και ΝΑΤΟ δεν έχουμε ε, δομή διοικητική που, θα, μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε κάτι τέτοιο και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε δυνάμεις και προσωπικό για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καμία ολοκληρωμένη διοικητική δομή επίσης. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν ε, τα ε, στοιχεία αυτά, να τα, τις διευκολύνσεις, με συγχωρείτε αυτές, να τις θέσουν ε, σε, στην διάθεση αυτού το οποίου θα ηγηθεί μια τέτοια επιχειρήση. Τα πάντα λοιπόν είναι στα χέρια και στον έλεγχο των κρατών μελών. Ε, είπα ότι εκπρόσωπος θα πρέπει να δει αν υπάρχει βούληση εκ μέρους των κρατών αυτό να αναλυφθεί μια τέτοια δέσμευση. Συζητούμε τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν επιτά. Επιτός θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισίες του καθενός και οι προσδοκίες του καθενός. Έτσι έχουν τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ενεργήσουμε. Αυτό το οποίο ε, θεωρείται ως ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε. Θα επανέλθω σε μία ή δύο εναλλακτικέ λύσεις τις οποίες εσείς αναφέρατε. Απλώς ήθελα ευθύς εξ αρχής να κάνω αυτό το γενικό σχόλιο. Κύριε Γκάλα, ρωτήσατε για θέματα σχεδιασμού και ποιο είναι υπεύθυνο στο στρατιωτικό επιτελείο και μαζί με το στρατιωτικό επιτελείο η διεύθυνση ε, διαχείρισης κρίσεων που είναι αρμόδια επί ε, της ουσίας και πρόκειται για μια ομαδική δουλειά και θα συνεχίσουμε ε, να ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Η υποστήριξη τώρα από την περιφέρεια. Υπάρχει εν μέρη, υπάρχει τοποθέτηση του Συνδέσμου του Αραβικού. Θα διαβάσατε βεβαίως ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε μαζί με τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Αφρικανική Ένωση να διαβουλευτεί. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα λάβουν χώρα αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα πρέπει να είναι καταπήγουσα συνεδρίαση. Ε, είμαι σχετικά βέβαιος ότι ο πρόεδρος Φαν Ρόμπαϊ θα ε, ερωτηθεί εδώ αύριο στο Κοινοβούλιο το θέμα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρυφτούμε πριν από την Αφρικανική Ένωση. Χρειαζόμαστε όμως αυτή την υποστήριξη από την περιφέρεια. Είναι προϋπόθεση αυτή προϋπόθεση του ΝΑΤΟ. Ξεκίνησατε στα γερμανικά να συνεχίσω και να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Μπράμνερ. Η εφαρμογή του εμπάρκο πρόκειται για τμήμα αυτού του prudent planning. Δηλαδή υπάρχει μια δυνατότητα, αν και θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι μια ε, δυνατή θέση δεν θα διέφερε πάρα πολύ, δεν θα απήχε πάρα πολύ από την ε, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Τώρα, ότι δεν θα γινόταν ε, με το εμπάργκο, θα γινόταν από τη θαλάσσια οδό. Έχουμε δηλαδή μια δυνατότητα μια θαλάσσια. Εξετάσαμε μάλλον τη δυνατότητα θαλάσσια αποστολή. Δεν ξέρουμε όμω τα αποτελέσματα και φυσικά χρειαζόμαστε και σχετική εντολή. η έννοια της προστασίας, της ευθύνης για προστασία, το γνωρίζουμε ασφαλώς, αλλά δεν είναι δεσμευτική αυτή, αυτό το σχέδιο, αυτή η ιδέα. Η εφαρμογή της έννοιας αυτής θα χρειαζόταν μια διαφορετική εντολή. Αυτό ασφαλώς ε, θα σήμαινε μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ που δεν έχει γίνει πλήρως. Δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμη. Δηλαδή, αναφέρατε και μία παράθεση από το Ίδρυμά μας. Θα μπορούσαμε να δώσουμε διαφορετικές ερμηνείες, αλλά δεν θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τόσο εύκολα εφαρμόσιμα. Για τα σχόλια τώρα του κυρίου Γκουαλτιέρη. Και μία άλλη ερώτηση για το πώς ε, γνωρίζουμε, τι γίνεται σε όλα τα μέρη της χώρης, χώρας. Έχουμε τις εικόνες από τους δορυφόρους που είναι αξιόπιστες αλλά όχι πλήρες. Και είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς, να εκτιμήσει την κατάσταση στη Βενγάζη, γύρω από τη Βενγάζη και εξαρτώμεθα κατά κάποιο τρόπο από τις εκθέσεις που αποστέλουμε κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε στείλει ερευνητικέ επιτροπές και στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη τις τελευταίες μέρες για να μας αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε επαφές με διάφορους φορείς επιτόπου. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ξέρουμε ότι συζητήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα της ενδεχόμενης αναγνώρισης του προσωρινού συμβουλίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι δεν ε, υπήρξε ομοφωνία. Θεωρείται ότι πρόκειται για έναν έγκυρο συνομιλητή. Συνομιλητής είναι και αυτή είναι η προσέγγισή μας. Εμείς σε επίπεδο συμβουλίου και με τους ε, συναδέλφους της CIS, της δύναμης που έχει και με την Λέδη Άστον, το συζητούμε αυτό το θέμα. Αλλά οι πληροφορίες που έχουμε είναι κατακαιρματισμένες ακόμη. Οι κυρώσεις, όπως σας είπα, εάν εφαρμοστεί το εμπάργκο, δεν θα είναι πολύ διαφορετική κατάσταση από ότι αν υπάρξει στρατιωτική επιχείρηση. Και βεβαίως σε επίπεδο ΝΑΤΟ το συζητώνται αυτά τα πράγματα και πρόκειται για μια δυναμική εξελισσόμενη. Συνεχίζουμε τη συζητήση με τα κράτη-μέλη και σήμερα το απόγευμα και σε επίπεδο ΝΑΤΟ σήμερα θα παρουσιαστούν και άλλα έγγραφα. Σύμφωνα με τα μέσα, επίσης, υπάρχει στη Λιβύη και πρόβλημα ε, ρευστού χρημάτων. Και μία από τις κυρώσεις θα ήταν να επιβληθούν και κάποιοι περιοριστικοί κανόνες σε επίπεδο χρηματοδοτικό και σε επίπεδο πίστης. Στον Μπαχρέιν τώρα τελικά. Για τον Μπαχρέιν. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης. Ξέρουμε ότι κάποια στρατεύματα από τη Σαουδική Άρα επίσης προσπαθούν να παρέμβουν για να υπερασπίσουν την κυβέρνηση. Και στην Ιεμένη υπάρχουν εξελίξεις. Όλες αυτές οι ενέργειες συνδέονται μεταξύ τους και πιστεύω ότι το θα συμβεί με τη Λιβύη τις επόμενες μέρες θα είναι αποφασιστικό για όλη την περιοχή. Έξι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ να είστε αρκετά σύντομοι και να επικεντρωθείτε σε ερωτήσεις. Από τις 11.30 ε, ήρθαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τη Λιβύη. Και τελικά ε, δαπανούμε το χρόνο σε μη επίγοντα θέματα. Κοιτάζω τα πρόσφατα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω τα ίδια κενά σλόγγαν, ε, τα οποία είναι αντιφατικά τα μεν ως προς τα δε. Οι δράσεις μας είναι κυρίως θέλουν να προστατεύσουν τους αμάχους. Ε, υπάρχουν όμως διάφοροι, ε, διάφορες πολιτικές προϋποθέσεις Ε, αν κάποιος διαφωνεί, δηλαδή κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά δεν υπάρχουν μέσα για να αναπτύξουμε κάποια δράση. Τα κράτη-μέλη, λέει, ετοιμάζονται για να ετοιμάσουν τη θέση, όχι να επιβάλλουν τη θέση, να ετοιμάσουν τη θέση. Τη θέσπιση μάλλον μία ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη, εάν το εγκρίνει το ΟΗΕ. Εύκολο δηλαδή. Δεν υπάρχουν σκεπτικισμοί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να εκφράσει η ΒΕΤΟ η Ρωσία ή η Κίνα. Μία αρκεί. Δηλαδή ένα βέτο αρκεί για να μην κάνουμε τίποτα. Το Κοινοβούλιο, λέει, ε, στεναρά ε, υποστηρίζει τις νόμιμες διεκδικήσεις του λιβικού λαού. Πραγματικά τις υποστηρίζουμε ή μόνο στεναρά τις υποστηρίζουμε. Για την ανθρωπιστική βοήθεια, λέει. Εξετάσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις χωρίς υπεφυλάξεις ή μόνο θεωρητικά εξετάσουμε τις ε, εναλλακτικέ λύσεις χωρίς να υπάρχει η μονο θεωρητικα εξετασουμε τις εναλλακτικες λυσεις βούληση για να τις εφαρμόσουμε. Τώρα για να τελειώσουμε. Τελειώνουμε γενικά με σλόγγαν. Ποτέ πια ε, λέμε αυτή τη στιγμή, που ο Καντάφη ε, καταλαμβάνει τη Βενγάζη και την, την εκαθαρίζει διώχνοντας χιλιάδες ανθρώπους. Τι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ πια. Τι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ πια. Πόσες φορές θα το επαναλάβουμε. Μετά την ε, Στρεμπρενίτσα, την Τζετσενία. Πότε, πόσες φορές πρέπει να ξαναπούμε ποτέ πια εις Το Συμβούλιο λέει ότι αυτό το προσωρινό ε, Συμβούλιο της Βενγκάζης θεωρείται ένας πολιτικός, λέει, συνομιλητής. Ενώ το καθεστώς του Καντάφη δεν είναι πια συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να έχει και πολιτικές συνέπειες όμως, ουσιαστικές συνέπειες. Αλλά μοιάζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απέναντί της δύο κυβερνήσεις. Η μία θεωρείται νόμιμη και αναγνωρισμένη, αυτή της Μπενγκάζης, ενώ η προηγούμενη είναι ήδη παράνομη και μη αναγνωρισμένη. Αυτή στην Τρίπολη δηλαδή. Και το Συμβούλιο λέει κάνει έκκληση να παρατηθεί η κυβέρνηση αυτή. Αλλά ο Καντάφη μας κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε απέναντί μας δύο κυβερνήσεις ταυτόχρονα. Έχουμε επίσης το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου που θα πρέπει να διασφαλίσει ε, την εθνική ακαιρεότητα και την ενότητα της Λιβύης ε, στη Βενγάζη και στο, στην Τρίπολη. Δηλαδή, και ο Καντάφη είναι ένας από αυτούς που θα εξασφαλίσουν αυτή την ενότητα. Μήπως είναι η ενσάρκωση του λαού του. Ε, επίσης, γίνεται έκκληση να διαφυλάξει την ειρήνη. Τι νόημα έχει αυτό όταν η Μπενγκάζη ήδη πολιορκείται. Και ετοιμαζόμαστε για πραγματικό πόλεμο εκεί πέρα, εντός ημερών. Ο Αραβικός Σύνδεσμος είναι μη ρεαλιστικός δηλαδή ή θεωρεί ότι ο συνταγματάρχης ε, Καντάφη είναι ένας ειρηνοποιός ο οποίος θα επιβάλλει την τάξη σε αυτό το τμήμα της Βόρειας Αφρικής. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να συγκρίνω την κατάσταση στην Πενγκάζη και την εξέγερση Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις, αλλά μου θυμίζει τη Βαρσοβία το 1944. Μου θυμίζει την εξεγερμένη Βαρσοβία, που έλεγε ελευθερία, και η οποία πολιορκήθηκε από τους Γερμανούς. Από το γερμανικό στραβό βομβαρδίστηκε, καταστράφηκε όταν ο Σοβιετικός στρατός έμεινε, έμεινε εβδομάδες πίσω πίσω από τον ποταμό Βιστούλα και περίμενε. Η ίδια κατάσταση είναι στη Λιβύη. Περιμένουμε τελειώσει η εξέγερση δηλαδή. Και εμείς δηλαδή, θα περιοριστούμε στην υποβολή συλληπιτηρίων. Ευχαριστώ κύριε Σαρλάκη. Μια σύντομη δήλωση. Και εγώ αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση από την έλλειψη αποφασιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά τα πρώτα, την πρώτη στιγμή μετά την κρίση. Και πιστεύω ότι υπάρχει αιμονή στις συζητήσεις ε, στο θέμα της χρήσης δύναμης. Η χρήση στρατιωτικών μέσων είναι μία από τις εναλλακτικέ λύσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή δεν έχει τίποτα ειδικό, το ιδιαίτερο να πει. Η, χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία είναι η ΕΠΑ. Αποφάσισαν να γίνουν ειρηνιστές, τώρα ανακάλυψαν το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Διεθνές Δίκαιο, και είπαν στον ΝΑΤΟ να κάνει αυτή τη σημαντική δήλωση. Τώρα εμείς θα πρέπει να διερευνήσουμε τις εναλλακτικέ λύσεις. Το να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση με πάρα πολλά θύματα ε, είναι μια δυνατότητα. Ε, το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν είναι τόσο εύκολο νομίζω, μερικοί. Αν γίνει σωστά, είναι ακόμα πιο δυνατό εργαλείο από μια στρατιωτική δράση. Αλλά πρέπει να γίνει με σοβαρό τρόπο. Πρέπει να γίνει σύμφωνα ε, με, ένα, με μια δέσμη τεχνικών κανόνων που μέχρι στιγμής δεν έχουμε διερευνήσει επαρκώς. το πάγωμα και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή κυβερνητικών αξιωματούχων δεν είναι καθόλου εύκολο στοιχείο. Υπάρχουν εμπειρίες. Ο ΙΕ έχει εμπειρία σε αυτό το τομέα και θα πρέπει να διερευνήσουμε αυτό το σημαντικό εργαλείο. Το δεύτερο εργαλείο που πρέπει να το κοιτάξουμε δεν είναι μόνο το εμπάργκο όπλων, αλλά η μείωση των όπλων. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, ε, υπάρχει ένα παράδοξος. παράδοξο. Χώρε που μέχρι χθε έδιναν εξοπλισμού στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή σήμερα ε, χρησιμοποιεί τα όπλα αυτά εναντίον των ε, υπερμάχων της δημοκρατίας. Και σήμερα ε, λένε πρέπει να σταματήσει η παράδοση όπλων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί πρόσφατα. Και μόνο στις έξι χώρες του κόλπου, στα πλαίσια της συνεργασίας του κόλπου, για το 2011 έχουν συμβάσεις για, για να λάβουν όπλα από δυτικές χώρες και από τη Ρωσία κτλ. αξίας 50 δις ευρώ. Μια και υπάρχει περίπτωση η κρίση αυτή να επεκταθεί και στη Σαουδική Αραβία και στον Μπαχρέν και τα λοιπά, στη Μέση Ανατολή δηλαδή, το παράδοξο είναι ότι αυτά τα όπλα θα, θα χρησιμοποιήσουν αυτέ οι χώρε. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί λοιπόν και να διερευνήσουμε εναλλακτικέ λύσει στην βίαιη χρήση στρατιωτικών μέσων, θα πρέπει να ζητήσουμε την αναστολή ε, των συμβάσεων αυτών για την παράδοση όπλων στις χώρες του κόλπου. Αυτό θα συνεισφέρει πολύ στην ειρήνη, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα είναι πολύ πιο σημαντικό από το σχέδιο Μάρσαλ που ετοιμαζόμαστε να εφαρμόσουμε. Υψούς, ε, δηλαδή 10 δισεκατομμύριων ευρώ. Μόνο αν μειώσουμε τους εξοπλισμούς κατά 50% θα μπορούσαμε να έχουμε για αυτή τη μεταβατική φάση της δημοκρατίας πολύ περισσότερους πόρους. Γιατί δεν διερευνούμε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, αντί να συνεχίσουμε με αυτές τις αιμονές που έχουμε για αυτή τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, για τη χρήση στρατιωτικών μέσων κτλ. Ευχαριστώ κύριο Λιζέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ποπόφσκι. Θα συμφωνήσω με αυτή τη μεγάλη την ομάδα των απογοητευμένων, γιατί πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλα ακράτη κράτη-μέλη κατηγορούν την Κριάστον, τη ΣΥΠΑ και τις διεθνείς οργανώσεις. Αναφέρθηκαν κάποια κίνητρα από τους συναδέλφους μου και ο κύριος Ποπόφσκι τοποθετήθηκε. Θα ήθελα όμως εγώ να κάνω μια γενική παρατήρηση για το κατά πόσο η κυρία Άστον συνειδητοποιεί ότι η τρέχουσα κατάσταση εκτιμάται από πολλούς πολιτικούς παρατηρητές ως ένα είδος ε, δοκιμασίας, όχι μόνο για τις προσωπικές της ικανότητες, αλλά και μια δοκιμασία για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη γιατί όπως φαίνεται υπάρχουν ε, θέματα επικοινωνίας μεταξύ της ΥΠΑ της ε, εκπροσώπου και των κρατών μελών. Τα κρατημέλη συμπεριφέρονται με πολύ διαφορετικό τρόπο και εμείς απέχουμε παρασάγκας από μία ε, κοινή, από ένα κοινό ψήφισμα και ίσως να υπάρχει και ένα θέμα επικοινωνίας με τα τρίτα κράτη τα οποία αντιδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική και δεν εννοώ τη ΣΥΠΑ. Είμαστε πολύ διστακτικοί, αλλά και τη Ρωσία. Από ιστορικής άποψης, η Ρωσία έχει και είχε πολιτικά συμφέροντα με την ε, Λιβύη και φυσικά σήμερα ε, τα, τα οικονομικά συμφέροντα είναι και αυτά πολύ σημαντικά και εδώ πέρα αναφέρομαι στο εμπόριο όπλων. Αν υπάρχουν διμερείς σχέσεις μεταξύ της κυρίας Άστον ε, και της Ρωσίας, πώς διαμορφώνονται. Merci, Monsieur Kirillov. Ευχαριστώ, κύριος Κυριλόφ. Γρήγορα σας παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, μία ερώτηση. Νομίζω ότι άκουσα ότι αποστέλλεται μία αποστολή στην Τρίπολη και στη Βεγγάζη. Τι θα κάνουν τα μέλη της. Θα έχουν με το καθεστώς του Καντάφη. Γενικά νομίζω ότι είναι αντιπαραγωγικό και νομίζω ότι πέσαν στην παγίδα τα μέσα ενημέρωση έστειλαν κάποιους στην Τρίπολη και εκδιώχθησαν όπως και κάποιοι δημοσιογράφοι που πήγαν από μόνοι τους και υπέστησαν κυρώσεις. Γιατί πάμε λοιπόν εκεί, τουλάχιστον από πολιτικής πλευράς έχουμε εκφράσει την θέση μας εμείς το καθεστώς. Και υπάρχει κάλυψη από κάποια μέσα που επειδή χειραγωγούνται από το καθεστώ Καντάφη δεν αποδίδουν την σωστή εικόνα της κατάστασης. Τι κάνουν λοιπόν. Δεύτερον, από όσον ξέρω δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πλοία στην περιοχή. Έχουν στείλει, ε, υπάρχουν αμερικανικά ε, αεροπλανοφόρα, αλλά δεν υπάρχει δική μας καμία τέτοιου δύναμη. Εάν η κατάσταση είναι σε τόσο κρίσιμη κατάσταση και όπως είπε ο κύριος Λανσμπέργκης θα αρχίσουν να υπάρχουν ε, μαζικοί βομβαρδισμοί πόνο λοιπόν, και κυρίως της Τρίπολης δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν να το επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι. Μιλούμε για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τέτοιους βομβαδισμούς. Τελευταία ερώτηση. δεν ε, παρακολουθούμε με πολύ επαγγελματικό τρόπο τι γίνεται. Παρακολουθούμε τι γίνεται μέσω των εικόνων που μας στείλουν οι δορυφόροι. Τι γίνεται ε, νοτίως και της ε, ε Τρίπολης, το νότιο μέρος της Λιβύης και εκεί υπάρχει εμπάργο. Τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Εάν επιβληθεί εμπάργο, επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι στη Βενγάζη. Διότι κατά την άποψή μου η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας στρέφεται κατά των αμάχων και του πληθυσμού. Ευχαριστώ κύριο Στράσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, δυστυχώς ε, θα πρέπει να συμφωνήσω με τα σχόλια που ανέφεραν μια μεγάλη δυσαρέσκεια για την παρουσίασή σας. Δυστυχώς αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Η έκθεσή σας, τα δηλώσεις σας, δυστυχώς καταδεικνύουν με απερίφραστη σαφήνεια πόσο αδύναμη και ανίκανη για ενέργειες και πόσο ανίκανη γενικότερα είναι η Ευρώπη σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Το πιο συγκεκριμένο στοιχείο στην παρουσίασή σας ήταν ότι κάποτε θα υπάρχει, θα, θα, θα λάβει χώρα μία ε, διάσκεψη κατεπίγουσα. Δεν είναι αυτό που περίμενε και περιμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης, κοιτώντας την προηγούμενη εβδομάδα, στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, οι πληροφορίες που λάβαμε όλοι μας ε, υποδείκνυαν ότι η μεταβατική κυβέρνηση αποτελούσε τελικό στόχο και ήταν σαφείς οι δηλώσεις που ακούσαμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πολύ καλή συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο αλλά και από τον Πρόεδρο Μπαρόσο και θυμάμαι αυτό που ανέφερε ότι θα πρέπει να φύγει ο δικτάτορας από τη Λιβύη. Τόσο σαφείς ήταν ε, οι δηλώσεις, το δήλωσε και ο Πρόεδρος Μπούζεκ Άρα γενικά υπήρξε ένας γενικότερος ε, σαφής όρος στον οποίο συμφώνησε όλη η Ευρώπη ότι συμφωνεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Μάλλον αυτό, ο, είχε τεθεί ο όρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Ε, συμφώνησε το, το Σαββατοκυριακό ο Αραβικός ε, Σύνδεσμος και τώρα περιμένω να ενεργήσει με σαφήνεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα μας λέτε, μα τον άτομα, ο Καταλαβαίνετε εσείς προσωπικά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αλλά σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τις πληροφορίες αυτές. Απευθύνω έκκληση. Είναι αυτονόητο. Και ο κόσμος που ήρθε και από τη μεταβατική κυβέρνηση και κάθισε μέσα στα έδρανα της Ολομέλης στο Στρασβούργο, μεταβιβάζουν τα μηνύματα αυτά. Το είπαν και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, το είπε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπαν ότι η Ευρώπη δεν είναι ουδέτερη, ότι στέκεται και υποστηρίζει την μεταβατική κυβέρνηση. Και ο κόσμος λοιπόν περιμένει μια αποφασιστικότητα. Μα και εγώ αυτό αναμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι. Και αυτό μου λείπει από την έκθεσή σας. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνετε και να επιβάλλετε μια ζώνη απαγόρευση πτήσεων, ναι, ότι θα πρέπει να επιβάλλετε μπάργκο Υπάρχουν πολλέ καλέ προτάσει. Αλλά αυτό που μου λείπει, αυτό που λείπει από την έκθεσή σα είναι μια θέληση, μια προθυμία διαμόρφωση τη κατάσταση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα ήθελα να υπάρχει. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να επανέλθουμε σε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Κυριλό, θα πω το εξή. Όντως στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ε, είχαμε τα αποτελέσματα μίας ε, αποστολής στην Τρίπολη. Για να μπορέσει κανείς να έρθει σε επαφή με τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27 ή όσων έχουν απομείνει, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο που περιμένει κανείς ε, ε, να έχει μετά από την επίσκεψη μιας αποστολής. Διότι κάτι τέτοιο μπορεί να εκλειφθεί και εάν ε, από τον Καντάφη ενδεχομένως σαν ε, υποστήριξη των ε, δράσεών του. Ελπίζω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο δεν θα επανελθεί. Και με τις νέες τεχνολογίες σήμερα τέτοιου είδους εκθέσεις μπορούμε να τις έχουμε και με τη βοήθεια του ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο κόσμος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την συζήτηση που έγινε και θα ήθελα να σας πω ότι θα υλοποιήσουμε όλες τις προσδοκίες. Αλλά ξέρετε σε ποιο πλαίσιο κινούμεθα. Αν πρέπει να συνάγουμε κάποια πορίσματα από την όλη κατάσταση, πράγμα το οποίο γίνεται, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διοπιστώσουμε ότι υπάρχουν κάποια περιορισμοί, κάποια όρια. Υπήρξαν πολλές προσδοκίες σε σχέση με την θέση σε ισχύ της νέας συνθήκης της Λισαβόνης. Κάποια πράγματα όμως δεν άλλαξαν. Οι κανόνες για την ε, ΚΕΠΑ δεν έχουν αλλάξει. Χρειαζόμαστε ομοφωνία. Τα μέσα που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για διαχείριση κρίσεων είναι μέσα και διευκολύνσεις των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να τα διαθέσει, εάν δεν το επιθυμεί. Και το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι κλειδί. Δεν μπορεί κανείς αν δεν έχει περαιτέρω εξουσιοδότη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να κάνει τίποτε περισσότερο, να προχωρήσει περισσότερο. υπήρξε μια ερώτηση για την επικοινωνία με τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να απαντήσω στα πολωνικά, αλλά ας απαντήσω αγγλικά. Μιλήσαμε με τους διάφορους συνομιλητές και τρίτες χώρες και με τους Ρώσους. Δύο φορές τις τελευταίες δέκα ημέρες και στη Γενέβη και χθες το βράδυ στο Παρίσι και με τον κύριο Λαυρόφ. Ξέρουμε ποια είναι η δική τους άποψη. και η επικοινωνία με τους Αμερικανούς είναι πάρα πολύ εκτεκταμένη και αυτό είναι πρόκληση και δοκιμή για όλους μας. Αλλά και με την καλύτερη θέληση εκ μέρου τη ΥΠΑ εκπροσώπου δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα γιατί έχουμε ακόμη στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας κάποια όρια μέσα στα οποία κινούμεθα. Ανέφερα προηγουμένως μια αποστολή και καταλαβαίνω τις επικρίσεις. Δεν ήταν υψηλού επίπεδου, δεν ήταν πολιτική και ο στόχος δεν ήταν να υπάρξουν συνομιλίες με την κυβέρνηση Καντάφη και δεν έγινε και κάτι τέτοιο εξάλλου. Ήταν αποστολή IAS για να μιλήσουν τα μέλη της αποστολής στην Τρίπολη με τους πρέσβεις μας, με συναδέλφους της ε, ΕΚΟ που ασχολούνται με θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κομισιό και ο στόχος του ταξιδιού στη Βενγκάζη ήταν να μιλήσουν επί τόπου με τα διάφορα άτομα, κυρίως και με μέλη του προσωρινού συμβουλίου για να δουν εκείνοι πώς ερμηνεύουν την όλη κατάσταση και την αξιολογούν. Χρησιμοποιούμε το κέντρο το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ξέρουμε τι συμβαίνει για να βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Μας αποστέλουν συνεχής εκθέσεις της εξέλιξης της κατάστασης σε όλη την ε, Βόρεια Αφρική αν θέλετε. Έγιναν επίσης ε, και κάποιες ερωτήσεις για τα μέσα, και τις διευκολύνσεις σε επίπεδο θάλασσας. Δεν κάνουμε εμείς ε, τίποτε. Ε, το Endeavour είναι εκεί και διάφορα άλλα αεροπλανοφόρα κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και στην ε, διάσκεψη των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο ανώτατος διοικητής είπε ότι προτίθεται να αναπτύξει κάποιες ναυτικές δυνάμεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε και να σχολιάσω καμία απόφαση του ΝΑΤΟ, γιατί δεν είμαι μέρος του ΝΑΤΟ. Υπάρχει όμως ε, ε, ναυτική παρουσία, όχι μόνο αμερικανική, στην περιοχή. Και βεβαίως θα μεταφέρω το μήνυμα της πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε. Και αυτό που είπατε φυσικά για την ε, ε, προθυμία και τη διάθεση διαμόρφωσης και την ικανότητα διαμόρφωσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τα μεταφέρω αυτά στην είπατη εκπρόσωπο που βρίσκεται ε, στο δρόμο της επιστροφής από την συνάντηση G8 στο Παρίσι που ουσιαστικά μετατράπηκε σε συνεδρίαση κατεπίγουσας ε, σημασίας, παρόλο που δεν είχε προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνειδητοποιούμε το γεγονό ότι η θέση σα δεν είναι εύκολη, αλλά νομίζω ότι ήταν απαραίτητο εμεί να σα μεταφέρουμε τα ερωτηματικά μα, τα σχόλιά μα, την απογοήτευσή μα, θα έλεγα επίση, όχι μόνο όσον αφορά την ε, ε, εφαρμογή κάποιας εναλλακτικής λύσης σε σχέση με κάποια άλλη. Αλλά από τη στιγμή που αναγνωρίζει το Συμβούλιο ότι θα πρέπει οι εναλλακτικές λύσεις όλες να τεθούν επιτάπητος, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε προς το παρόν. Παρά το γεγονός ότι είναι η εντολή δύσκολη, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν Αύριο ο πρόεδρος Βον Ρόμποϊ θα λάβει το λόγο στη διάσκεψη των ε, Προέδρων, ανοιχτή συνεδρίαση στη 1.30 για όλους και την επόμενη εβδομάδα η κυρία η Λέιδη Άστον την Τρίτη θα λάβει το λόγο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την επαύριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και την παρέμβασή σας.